Α, ήρθες για να μείνεις. Πάρα πολύ ωραία. Καλά το σκέφτηκες. Ας αφήσουμε όμως τα αστιάκια να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν υπάρχουν προτάσεις τροποποίησης, εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ως ε, ήθιστε. Σας ε, δίνονται τα πρακτικά τα οποία στο τέλος ε, της συνεδρίασης και αν δεν έχουν υπάρξει κάποιες τροποποιήσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Έγκριση σχεδίου χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων της Επιτροπής μας για τον επόμενο χρόνο. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλες τις απαιτήσεις, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των συναδέλφων. Έχουμε βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα, έτσι το πρώτο σχέδιο που μας δίνει το κοινοβούλιο, βλέπουμε, ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε έτσι σημαντικά προβλήματα, επικαλύψεις συνεδριάσεών μας ε, με συνεδριάσεις άλλων επιτροπών. Ε, ό,τι καλύτερο μπορέσαμε το κάναμε και θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα είναι καλό και να το εγκρίνουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αν δεν υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί εγκεκριμένο να σας πω ότι εντωμεταξύ συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ε, ε, πέρα από, την, το ταξίδι της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, ε, προσεκλήθη στην Ελλάδα επίσης τον ε, Σεπτέμβριο και είχα την δυνατότητα να συναντήσω τον ε, Υπουργό κύριο χοίδη υπεύθυνο μεταξύ άλλων και της ανάπτυξης αλλά και της περιφερειακής πολιτικής ο οποίος μάλιστα αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να παραστεί στην συνεδρίασή μας του Νοεμβρίου έτσι ώστε να αναφερθεί στις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα έτσι ώστε ε, να ε, χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα και να αναπτύξει την ε, ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. και αυτές οι αποφάσεις ε, ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις των συντονιστών της 22ης ε, Σεπτεμβρίου. Έγιναν συζητήσεις ε, βάσει του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου έλαβε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για τον τροποποιητικό δηλαδή κανονισμό. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ε, η διαδικασία επήγει ε, και επομένως οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η Πρόεδρος θα είναι υπεύθυνη για την σύνταξη γνωμοδότησης για, αυτές τις, για αυτούς τους κανονισμούς. Επίσης, Βάσει της απόφασης των συντονιστών, ε, η εισηγήτρια θα πρέπει να κάνει διάφορες ε, διερευνητικές ε, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και επίσης να συντάξει το προσχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης, βάσει πάντα των αποφάσεων των συντονιστών, ε, προτείνομαι να γίνει τη 14η, 14η Νοεμβρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας έτσι ώστε στην επόμενη Ολομέλεια ε, να ε, περάσει το θέμα αυτό. Επίσης συστήνουν προς την, μάλλον όχι, αποφάσισαν οι συντονιστές να αποσυρθεί το αίτημα που είχε υποβληθεί για μια ε, ίδιας ε, πρωτοβουλίας έκθεση για, τις ε, δημόσι... για τους δημόσιους διαγωνισμούς βάσει πληροφοριών που είχαμε ότι θα επανακάμψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τροποποίηση των προτάσεων σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς και επομένως θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτήν την γνωμοδότηση νομοθετικού περιεχομένου. Τελευταία ανακοίνωση για σήμερα. Ε, ο Κριστιαν Σοπέν που ήταν ε, εδώ από την αρχή της ε, θητείας, αλλά που είναι όμως παλιό, πολύ παλιό μέλος, 37 χρόνια υπηρεσίας έχει στις στις ε, ευρωπαϊκές ε, ε, υπηρεσίες. Επομένως είναι πραγματικά ένας θησαυρός που θα τον χάσουμε διότι συνταξιοδοτείται. Και αν μου επιτρέπετε εξ ονόματος όλων μας, μια και είναι η τελευταία φορά που θα είναι μαζί μας, Εκτός και αν θέλεις να έρχεσαι βέβαια όποτε θέλεις και να μας παρακολουθείς, είναι η τελευταία επίσημη ε, φορά που θα ε, παραστεί στην συνεδρίασή μας και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ε, προσπάθεια που έχει καταλάβει, καταβάλει, συγγνώμη, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα. And now, if you allow me, I will spare listening to the nightmares we are going through to, get replacement also. Because... Καλά, τώρα να μην συζητήσουμε τον εφιάλτη της ε, αντικατάστασης του Κριστιανού, γιατί οι διαδικασίες στο Κοινοβούλιο έχουν γίνει τόσο περίπλοκες που είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο ε, να ε, βρούμε κάποιον αντικαταστάτη αρκετά γρήγορα. Μιγέλ προσπαθεί όμως να κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Φτάνουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως που αφορά σχέδιο έκθεσης για το οποίο είμαι εισηγήτρια σχετικά με την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στα Κανάρια νησιά. Πρέπει να σας πω ότι το βασίλειο της Ισπανίας ζήτησε εξ ονόματος των αρχών των Καναρίων νήσων, που είναι αυτόνομη περιοχή, ζήτησε λοιπόν την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου ε, για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα κατά την εισαγωγή τους στα Κανάρια νησιά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τοπική ανάπτυξη, καθώς επίσης η διευκόλυνση κάποιων μικρομεσαίων τοπικών ε, παραγόντων και έτσι ώστε να βελτιωθεί και η ανταγωνιστική θέση της οικονομίας των Καναρίων νήσων. Επιβεβαιώνεται ότι η απόφαση δεν θα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού μια και ε, εστιάζεται περισσότερο στην στήριξη της τοπικής ε, ανάπτυξης ε, και, την ανάπτυξη, και στην ανάπτυξη των τοπικών φορέων και έχει επομένως συγκεκριμένη τοπική εμβέλεια. Προτείνω ε, λοιπόν να προχωρήσουμε με υποβολή τροπολογιών βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας ε, βάσει του άρθρου, δυνάμει μάλλον του άρθρου 46. Ε, Και επομένως να μην υπάρξουν τροπολογίες επί της προτάσεως αυτής που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεχτείτε λοιπόν την απλουστευμένη διαδικασία, δυνάμει του άρθρου 46 είπαμε, τότε ε, πριν από το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμα όλα και θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Um Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με αυτό ε, που προτείνεται, λέει ο κύριος Τεσέρα. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπατε ιδιαίτερα επί της ουσίας της πρότασης περί αυτού πρόκειται ενίσχυση ε, της οικονομίας των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, όπως είναι οι Κανάριες νήσι. Ε, αντίστοιχη πρόταση εγκρίθηκε για τη Μαδέρα και τις Ασόρες πέρσι τον Οκτώβριο. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα μέσα ε, πρέπει να έχουν και πρακτικά αποτελέσματα. Και κατά τύχη, πριν από δύο εβδομάδες, έλαβα ένα email που μου έστειλε επιχείρηση των Αζωρών, η οποία εξέφραζε παράπονα. Προσπάθησαν πριν από δύο μήνες να εισάγουν ένα μηχάνημα, ραπτική συγκεκριμένα, που τους χρησιμεύει για την εμπορική τους δραστηριότητα. Και είναι μια εταιρεία που εδρεύει στις Αζόρες, όπως σας είπα, και ε, φτιάχνει πανιά για καράβια. Και ήθελα λοιπόν να εισαγάγει αυτό το μηχάνημα που τους χρειάζεται και είναι και στο παράρτημα του κανονισμού που εγκρίθηκε πέρσι τον Οκτώβριο. Και ήρθε λοιπόν το τελωνίο των Αζωρών και τους είπε ότι δεν γνωρίζουν αυτό το κανονισμό. Και ήρθαν σε επαφή ε, και με το τελωνίο της Μαδέρας, το οποίο επίσης δήλωσε άγνοια του κανονισμού και τελικά η εταιρεία χρειάστηκε να πληρώσει το δασμό κανονικά για να εισαγάγει το μηχάνημα. Τι εννοώ, γιατί τα λέω όλα αυτά. Δεν έχει κανένα νόημα η δική μας δουλειά ε, υπέρ των ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, γιατί ε, εάν στη συνέχεια δεν ενημερώνονται οι υπηρεσίες και δεν τις υλοποιούν τις αποφάσεις, εγώ ήδη έχω κάνει μια γραπτή ερώτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή και ρώτησα αν έχουν κάνει διαβήματα Στι εθνικέ αρχές για να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Ορίζει ο κανονισμός ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, δημοσιεύουν και να γνωστοποιούν τα μέτρα αυτά. Ελπίζω αυτά που συνέβησαν στη Μαδέρα και τις Αζόρες να μην επαναληφθούν στα Κανάρια νησιά. Γιατί αλλιώς τι να το κάνουμε, να θεσπίζουμε νομοθεσία και τελικά να μην εφαρμόζεται και να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι επιχειρήσεις, είναι οι πολίτες, είναι ο κόσμος. Και αν υπάρχει κάποια ολιγορία ή αδράνεια από πλευράς των κρατών μελών ή των αρμοδίων αρχών, σε επίπεδο κρατών μελών, τότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε να τα διαβιβάσετε αυτά αρμοδίως και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στις εθνικές αρχές για να ε, δίνουν λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτά. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κανείς. Ή κάποιος από τους συναδέλφους ε, ε, θέλει να σχολιάσει, αλλά βεβαίως όλοι νομίζω ότι ζητάμε ε, να ε, κοινοποιηθούν στις διαφερόμενες αρχές άμεσα οι αποφάσεις έτσι ώστε πραγματικά η τοπική κοινωνία και η τοπική εμπορική κοινότητα <clears throat> να ωφεληθεί από αυτές τις προσωρινές αναστολές Θέλετε να εξηγήσετε κάτι, υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να επιβεβαιώσει τη δέσμευση τη ιδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πληροφορία αυτή πραγματικά μας εκπλήσει γιατί υπάρχει κανονισμός. Ο κανονισμός αυτός βεβαίως ε, εφαρμόζεται άμεσα ε, στα κράτη-μέλη γενικότερα, πολλό δε μάλλον ε, σε τις αφορόμενες περιοχές. Όσον αφορά το αίτημα, το, το ζήτημα μάλλον στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Βουλευτής, οπωσδήποτε ε, θα, και στην ερώτηση που υπέβαλε, οπωσδήποτε ε, θα με άμεσα. Ωραία. Πρόεδρος. Ε, επομένως ευελπιστούμε ότι δεν θα ξανά συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα θα ψηφίσουμε το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή μας. Α, συγγνώμη. Έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου ένα σύντομο σχόλιο, έτσι μια σκέψη που θέλω να προσθέσω σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Μαδέρα. Κατανοώ την αγωνία του, αλλά οι Ισπανικές αρχές εμπροκειμένου μετά από αίτημα των αρχών των Καναρίων νησιών ζητούν οι ίδιες οι αρχές να καταργηθεί ο τελωνιακός δασμός για να προσταθεί ο προστατευτεί ο βιομηχανικό κλάδο ο συγκεκριμένος που θέλει και συγκεκριμένα μέτρα και τα έχει ανάγκη και να προστατευτεί η οικονομία, η ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών που είναι τα Κανάρια αλλά και άλλα νησιά και είναι απολύτω απαραίτητο αυτό και για την Επιτροπή μα. Γι' αυτό χαίρομαι που η συγγήτρια συμφώνησε με τον κανονισμό αυτό και προτείνει να γίνει χωρίς τροπολογίες η έγκρισή του από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση ως το τέλος... Α, όχι, δεν, δεν ψηφίσουμε, λέει η κυρία Χούμπνερ. Ναι, γιατί είναι βάση του 46. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Ουσιαστικά τα σημεία 6 και 7 συνδέονται. Αν θυμάστε, σας το προανήγγυλα στο πλαίσιο των αποφάσεων των συντονιστών. Πρόκειται για αποφάσει τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δύο διαφορετικές αποφάσεις, δύο διαφορετικές διαδικασίες και δύο εκθέσεις. Οπότε, Ξεκινώ με το, σημείο 6. Η στρατηγική φυσικά έχει ήδη από του συντονιστέ, οπότε εντάχει σα ενημερώνω πριν ζητήσω από την Κομισιόν να λάβει το λόγο ότι ο λόγο κανονισμό είναι η ανταπόκριση μα στην κρίση και δι σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, τα οποία πλήττονται όλος ιδιαίτερος από την κρίση. Στον ελόγω κανονισμό και βάσει της υπόφασης των συντονιστών έγιναν ήδη πρώτες επαφές και ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Τις τελευταίες εβδομάδες ανταλλάξαμε απόψεις, πληροφορίες και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ανδέως τις θέσεις του Συμβουλίου Υπουργών, της Κομισιόν κλπ. Και να τις με τις δικές μας. Ο χρόνος πιέζει βεβαίως πάρα πολύ. Αν θέλουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση των συντονιστών, δηλαδή να προχωρήσουμε με μία και μόνη ανάγνωση, πρέπει να συντονίσουμε όσο γίνεται τις επιμέρους θέσεις, κυρίως μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων. Περιμένουμε από την Κομισιόν να μας δώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όσον αφορά δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις όλων αυτών των προτάσεων. Αυτό στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας η οποία σε, κανένα όργανο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ίσως έχει ολοκληρωθεί στην Κομισιόν, αλλά όχι στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που ακόμη συζητούμε τις προτάσεις. Γι' αυτό ακριβώ και δεν υποβάλλω σήμερα σχέδιο έκθεσης με τροπολογίες, όμως το επεξημενικό σημείωμα το οποίο σας έχω στείλει, Ευχαριστώ την προσοχή σας στους τομείς στους οποίους ε, χρειάζεται το κείμενο να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί ως προς το αρχικό δηλαδή κείμενο της Κομισιόν. Στόχος αυτών των τροπολογιών εντάχει είναι να κάνουμε κάτι για τις ε, ιδιαίτερες πληττόμενες χώρες μέσω της προσωρινής αύξησης της μέγιστης χρηματοδότησης συγχρηματοδότησης, αν θέλετε. Αυξάνουμε λοιπόν τα ποσοστά, χωρίς όμως να τροποποιούμε το συνολικό ποσό σε απόλυτες τιμές στο πλαίσιο της συνοχής για τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Οι χώρες που θα λάβουν βοήθεια συμπεριλαμβάνουν τις χώρες οι οποίε σήμερα συμμετέχουν στα προγράμματα μακροοικονομικής υποστήριξη Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία. Η πρόταση είναι αντικείμενο της ε, συνήθω νομοθετική διαδικασία, Οπότε στη φάση αυτή θα ζητήσω από τον Ρούντολφ Νίσλερ, τον διευθυντή αρμόδιο Διευθυντή Πολιτική Συντονισμού τη Ρίτζιο, της ε, γενική Διεύθυνσης Ρίτζιο, να μα ε, ενημερώσει εν συντομία. Και αν έχετε καλοσύνη κύριε Νίσλερ, μπορεί να έχουμε και ερωτήσει για εσά για να καταλάβουμε τη συλλογιστική που διέπει αυτέ τι αποφάσει. Προ το τέλο, μπορεί να πω και εγώ δύο λόγια πλέον σχετικά με τι τροπολογίε, αλλά ε, σας δίνω το λόγο, κύριε Νίσλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω εν συντομία να παρουσιάσω τα κυρία σημεία αυτής της πρότασης. Ο λόγος ύπαρξης αυτής της πρότασης είναι οι δύο, τα δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια το, πριν το καλοκαίρι, όπου τονίστηκε η ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τη συνέργεια μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των δανειακών διευκολύνσεων που έχουν λάβει ορισμένε χώρε. Στι 21 Ιουλίου, στις ε, διακήρυξει του Συμβουλίου, για την Ευρωζώνη, σουλιάστηκε κυρίως η κατάσταση της Ελλάδας. Και ζητήθηκε το μέτρο αυτό, δηλαδή της προσωρινής αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης για την Ελλάδα και για κάποιες άλλες χώρες. Η Κομισιόν προσπάθησε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα αυτό του Συμβουλίου και την του υπέβαλε πρόταση για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό δηλαδή που διαβάζετε εδώ μπροστά σας αφορά βέβαια στο Ταμείο Συνοχής η FSF και Ταμείο Συνοχής, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις, ταυτόσιμες προτάσεις για το Ταμείο και για το ΕΤΠΑ. Ο κύριος στόχος μας, εν προκειμένου, είναι υπό τις εξαιρετικές αυτές περιστάσεις της κρίσης να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες δίνουν μεγάλο αγώνα για να αντιμετωπίσουν το βάρος της χρηματοδότησης για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εκεί δηλαδή βοηθούμε τα συγκεκριμένα έργα με υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Η κεντρική ιδέα είναι πολύ απλή. Το σύνθεσ ποσοστό το αυξάνουμε κατά 10 ποσοστίες μονάδες. Η πρόταση, όπως είπε και η κυρία Χούμπνερ, αφορά αποκλειστικά τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και λαμβάνουν χρηματοδότηση βάσει των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Δηλαδή το EFSF εντός Ευρωζώνης και τους άλλους μηχανισμούς εκτός Ευρωζώνης. Με βάση αυτά λοιπόν όλες οι χώρες πρέπει να αντιμετωπιστούν επίσης όλες. Η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά την, την περίοδο επιλεξιμότητας. Η είσοδος της κάθε χώρας στο μηχανισμό αυτών στην πρόταση αυτή είναι και η ημερομηνία Έναρξη τη επιλεξιμότητας για το αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης. Και το τέλος, η εκπνοή αυτού του μέτρου, είναι και η ημερομηνία εξόδου από τους μηχανισμούς στήριξης. Όταν δηλαδή οι χώρε αυτέ θα επανέλθουν στην προτεραιά κατάσταση, τότε δηλαδή θα επανισχύσουν και τα συνήθη ποσοστά συγχρηματοδότηση. Το πράξαμε αυτό, ώστε από τεχνικής απόψεως η πρόταση να είναι απλή. για να μπορέσουμε η δράση μας να έχει άμεσο αποτέλεσμα όσον αφορά τις χρηματικές μεταφορές, τις μεταφορές κονδυλίων προς τις χώρες αυτές. Το καλό είναι ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί από τώρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε δηλαδή τίποτα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ταμεία αυτή τη στιγμή. Η εφαρμογή δηλαδή είναι, αν θέλετε, αυτόματη από τη στιγμή που η χώρα είναι ούτως ή άλλως επιλέξιμη βάσει του συγκεκριμένου κανονισμού. Τα επιπλέον κονδύλια δηλαδή θα χορηγηθούν, θα μεταφερθούν βάσει του κείμενου μηχανισμού, των κειμένων διαδικασιών. Ακούστηκε και η εξή πρόταση, το κράτος μέλος να ζητήσει επισήμως να επωφεληθεί από το συγκεκριμένο μέτρο στο πλαίσιο του κανονισμού και αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιήσει και η Κομισιόν ως αιτιολόγηση της αποφασής της. Όταν είπα ότι πήραμε μια γενναία απόφαση, ε, εννοώ ότι αφήνουμε τα προγράμματα συνεργασία ε, όπου εμπλέκονται και άλλα κρατημέλη, γιατί αυτό θα περιέπλεκε την κατάσταση και θα αλλίωνε και τα ποσά τα οποία θα πήγαιναν στη συγκεκριμένη χώρα κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γι' αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με τα μεγάλα προγράμματα. Δηλώνω επίση ότι δεν υπάρχει επίπτωση στον προπολογισμό. Απλώς αυξάνουμε κατά 10 ποσοστές μονάδες τη συγχρηματοδότηση. Άρα κάποια κονδύλια απλώ θα καταβληθούν νωρίτερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, για την καταβολή κονδυλίων του 12 δεν υπάρχει ανάγκη πλέον πιστώσεων, έγκριση πλέον πιστώσεων για να καλυφθούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Η Κομισιόν με την πρότασή της δεν προβλέπει και την ημερομηνία λήξη, διότι ούτως ή άλλω η αλλω η ενίσχυσης καθορίζεται από απόφαση του Συμβουλίου για την εκάστοτε χώρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτομάτως υπάρχει και ημερομηνία λήξη. Αυτό το συζητήσαμε στο Συμβούλιο, αλλά κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται. Έχει μεγάλη σημασία προκειμένου και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό ξεχωριστά είναι ότι ο μηχανισμός που προτείνουμε απαιτεί αναδρομική εφαρμογή. Ο στόχος είναι όταν τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι διατάξεις, το κράτος μέλος, το οποίο συμμετέχει σε πρόγραμμα στήριξης και το οποίο έχει υποβάλει αιτήσει κάλυψη δαπανών να μπορεί να επικαλεστεί την νέα διάταξη από τη στιγμή που ξεκίνησε ένα έργο ω την πρώτη πληρωμή. Έτσι, έχουμε την δυνατότητα να μεταφέρουμε στο συγκεκριμένο κρατός μέλος σημαντικά μεγαλύτερα ποσά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, οι σχετικέ διατάξεις πρέπει να καλύπτουν και αυτή το ενδεχόμενο καθώς και το 2010. Μίλαμε λοιπόν για 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ εδώ σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις των κρατών μελών. Όσον αφορά τις εμπλεκόμενες πληρωμές αλλά και τις μελλοντικέ, για τις οποίες δηλαδή θα ισχύσει ακριβώ το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Ως τώρα συζητήσει στο Συμβούλιο περιστρέφησαν γύρω από δύο κυρία ζητήματα και ο συνάδελφός μου από την Προεδρία από το Συμβούλιο με συγχωρείτε είναι εδώ για να σας πει περισσότερα αν χρειαστεί. Γύρω λοιπόν από τα εξή θέματα. Πρέπει η αναδρομικότητα, ο αναδρομικός χαρακτήρας να περιοριστεί και ενδεχομένω να προσθεθεί και μια και η πρόληψη λήξης του μέτρου. Όπως επίσης και το ποιε είναι οι χώρε που πρέπει να είναι επιλέξιμε. Αυτό βεβαίω θα σήμαινε ότι πρέπει να προβλέψουμε ρητό ποιε είναι οι χώρε για τι οποίε μπορεί να ισχύσει αυτή, αυτή η τροποποίηση, εκτό από αυτέ που συμμετέχουν ήδη στο μέτρο. Τώρα, όσον αφορά τον ρόλο τη Κομισιόν στην διαδικασία, για εμά, το σημαντικό είναι ότι η Κομισιόν θα εξετάσει ευμενώς τα αιτήματα των κρατομελών να αποφεληθούν από την τροποποίηση. Η Κομισιόν επίση θα αξιολογήσει και τη σχετική δικαιολόγηση. Αυτό το οποίο από την άλλη μεριά δεν θέλουμε να κάνουμε και δεν θα δεχθούμε είναι να δημιουργήσουμε μια επιπλέον διαδικασία βάσει τη οποία στο πλαίσιο τη οποία, μια Κομισιόν Κομισιόν θα κρίνει κατά περίπτωση εάν μπορεί να υποφεληθεί μια χώρα ή όχι. Εμεί πιστεύουμε λοιπόν αντιθέτω ότι η απόφαση του Συμβουλίου να εντάξει κάποιε χώρε αυτόν τον κανονισμό βάσει τη τροπή, αυτό θα είναι επαρκέ για την δρομολόγηση, για την κινητοποίηση του μηχανισμού, τη διαδικασία. Πρόκειται λοιπόν για αυτόματη εφαρμογή, αν θέλετε. Αυτό επιθυμεί η Κομισιόν για να μην προκύψουν και καθυστερήσει στην διάθεση τη επιπλέον στήριξης που προβλέπει ο κανονισμός. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να βοηθήσω εσά το Συμβούλιο, είμαι στη διάθεσή σας. Προσβλέπω στη συνεργασία μας τις επόμενε εβδομάδε. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να προχωρήσει αυτή η πρόταση. Οπότε, επαναλαμβάνω ότι είμαι στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μιλήσει αυτή τη στιγμή από την Προεδρία για να διευκρινίσει τίποτα το Συμβούλιο. Ο Ντίκ Πιόρ είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό εξ ονόμα της Πολωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω ότι ε, χειριζόμαστε αυτές τις τροπολογίε και τις τροποποίησεις μάλλον ε, ως ε, μέγιστη προτεραιότητα. Μέχρι στιγμής είχαμε πέντε ε, συναντήσεις, συνεδριάσεις στο Συμβούλιο, στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας και φαίνεται ότι θα συμφωνήσουμε για τις δύο τροποποίησεις. Διαφαίνεται αυτή η προοπτική, δεν είναι εύκολο. Αυτό το τελευταίο που ανέφερε ο Ρούντοφ Νίσλερ για την τελευταία τροποποίηση, αλλά φαίνεται ότι ε, έχει επιτελεστεί σημαντική και ουσιαστική πρόοδος. Προσβλέπουμε σε ολοκλήρωση των εργασιών στην ομάδα εργασίας μας, προσεχώς, θα σας παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα των εργασιών μας ε, εφόσον ε, προηγουμένως παρουσιαστεί στο κόρε πέρσι τη μονάδα μόνιμα αντιπροσώπων. Ευχαριστώ, Ραμόν. Να, ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Μανιάσκου, ε, διάβου, άκουσα προσεκτικά τα όσα είπε ο κύριος Νίσλερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθεί το συντομότερο ε, έκθεση αυτή έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που πλήττονται περισσότερο από την κρίση να έχουν την οικονομική υποστήριξη που χρειάζονται για να συνεχίσουν ε, τα προγράμματα και τα έργα. έχει μειωθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα πρέπει να πληγούν επιπλέον οι χώρες αυτές, οι οποίες είναι και αλλιώς αναγκασμένες να κάνουν μεγάλες οικονομίες. Είναι γνωστό ότι τα έργα αυτά θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα, θα εξασφαλίσουν διατήρηση των θέσεων εργασίας και θα τονώσουν την οικονομία. Και ταυτόχρονα ε, θα είναι και ένα μέσο καταπολέμησης της ε, ανεργίας. Είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών να αξιοποιούν όσο γίνεται περισσότερο ε, τα κονδύλια αυτά και να το εξασφαλίσουμε εμείς, να πιάνουν πραγματικά τόπο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια αυτά από τις πέντε χώρες το έτος 2010 οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Το 2010 τι έκαναν. Γιατί χρησιμοποιήσαμε αυτή την ευκαιρία, αξιοποιήσαμε αυτή την ευκαιρία εμείς να στηρίξουμε τις χώρες αυτές, αλλά θέλουμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Καλούμαστε τώρα να πάρουμε και άλλες τέτοιες αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι οι ε, κυβερνήσεις των κρατών αυτών αντιλαμβάνονται την ευθύνη που τις βαραίνει και χρησιμοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα κονδύλια. Και επίσης ε, θα ήθελα να μάθω, θα ήταν ενδιαφέρον αν υπάρχει ήδη κάποια αξιολόγηση σχετικά. Για να μην είναι στο βρόντο η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννα yes, I think that... Ευχαριστώ Γιάννα Ολμπριχτ. Έχω μερικά σχόλια και μία ερώτηση. Διότι καταρχάς υποστηρίζω την ιδέα της ε, τροποποίηση Είναι πολιτικό το μήνυμα και πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά ωραία. Αλλά μερικά σχόλια. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει, πιστεύω, ε, την απόφαση του Ιουνίου ότι η πολιτική συνοχής και τα μέσα της πολιτικής ε, συνοχή θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της κρίσης και σήμερα και αύριο. Αν αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά και όχι τελείως περιθωριακά αυτό το μέτρο. Χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία στα μέσα και για το μέλλον. Δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σαφείς στον ορισμό μας ότι αυτό το μέτρο είναι προσωρινό. Προσωρινό και όχι ένα νέο στοιχείο. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε και στους νέους κανονισμούς την κατάσταση, γιατί οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να είναι πολύ σαφείς. Έχουμε τη σημερινή εμπειρία και δεν μπορούμε να εργαστούμε με την ίδια αδράνεια του παρελθόντος στο νέο κανονισμό θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή για να γίνει κάτι στο μέλλον. Δηλαδή, στο νέο κανονισμό θα πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο αντίστοιχο. Και μια ερώτηση, με τις συνέπειες τι γίνεται. Δηλαδή, τα πάντα έχουν συνέπειες στη ζωή. Εάν έχουμε τώρα την προκαταβολή, ε, αυτό το έμπρο στο βαρές ε, ε, στο σύστημα, θα υπάρχουν συνέπειες στις χώρες αυτές του χρόνου. Και ποιες θα είναι αυτές, λιγότερα έργα ή χαμηλότερη συγχρηματοδότηση. Διότι, και το είπατε επανειλημμένα, τα χρήματα δεν είναι καινούρια επιπλέον, από κάπου τα παίρνουμε, δηλαδή από τα επόμενα έτη, ωραία. Και τα καταβάλουμε τώρα, προκαταβολικά, άρα του χρόνου θα είναι λιγότερα τα χρήματα αυτά, έτσι δεν είναι για να βγαίνει το άθροισμα τελικά μηδενικό. Λοιπόν, ποιε θα είναι οι συνέπειε, θα είναι λιγότερα τα έργα μεθαύριο που δεν θα έχουμε χρήματα ή θα είναι χαμηλότερη η χρηματοδότηση, για να ξέρουμε πραγματικά τι αποφασίζουμε και τι κάνουμε. Βεβαίω, ε, συμφωνούμε επί τη αρχή και με την ιδέα. Και μια πολύ μικρή ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Δεν γνωρίζουμε όλοι τι είναι sunset clause, δηλαδή ρήτρα λήξη, ισχύω ή ρήτρα εκνοή Θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Αγκουράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω να πω το εξή. Καταρχήν εκ πρώτη όψεω, φυσικά φαίνεται ότι αυτό το μέτρο μπορεί να βοηθήσει τι χώρε, οι οποίε αντιμετωπίζουν ε, τα γνωστά προβλήματα τη κρίση. Κατά τη γνώμη αυτή είναι όμως η όψη ε, των πραγμάτων και όχι η ουσία, αν κρίνω από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το πρώτο ερώτημα που έχω να θέσω είναι το εξής. Είναι προφανές ότι για την κρίση μεγάλο μέρος ευθύνη έχουν και τα προγράμματα τα οποία είχαν οι χώρες μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα αν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κρίσης θα χρειαστεί να βάλει ένα ερώτημα και ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων που να αντιμετωπίσουν την κρίση και όχι να την οξύνουν. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, το αντίθετο. Τα προγράμματα συνεχίζονται. Δεύτερον, στην περίπτωση της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, όταν ανακοινώθηκε αυτή η πρόθεση για την μείωση της εθνικής συμμετοχής στα κοινοτικά προγράμματα, υπόθηκε ότι αυτό γίνεται παράλληλα και με την περικοπή μεγάλου αριθμού κοινοτικών προγραμμάτων με το επιχείρημα της χαμηλής απορροφητικότητας. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αυτό το κριτήριο θα παίξει κάποιο ρόλο στο μέλλον. Τρίτο ζήτημα αφορά το θέμα των μεγάλων περικοπών που γίνονται αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους και στους δημόσιους υπάλληλους στη χώρα μου. Πρέπει να ξέρετε κυρία Πρόεδρε ότι έχουν αποφασιστεί περικοπές στους δημόσιους υπαλλήλους μέχρι και το 40%. Αυτό αφορά τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τα κοινωνικά προγράμματα, για το ΕΣΠΑ, για την απορρόφηση, για τα έργα και καταλαβαίνετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες μάλλον τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Κλείνοντας, πολύ φοβάμαι ότι μείωση εθνικής συμμετοχής, μεγάλη μείωση των προγραμμάτων, στην πράξη σημαίνει ότι κάποιοι οι οποίοι κερδίζαν μέχρι τώρα από την κρίση θα κερδίσουν ακόμα περισσότερα διότι είναι προφανέ λιγότερα προγράμματα, περισσότερα χρήματα, κάποιοι που ήδη είναι μες στα προγράμματα θα κερδίζουν περισσότερα και μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού θα υποφέρει ακόμα πιο πολύ. Άρα όξιση της κρίση. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω βεβαίως ε, στο βάρος της κρίσης που διανύουμε και το οποίο φυσικά ξεπερνά τα διαρθρωτικά ταμεία και τη χρηματοδότησή τους, αλλά ε, πρέπει να ενεργήσουμε σαν αλληλέγγυοι Ευρωπαίοι ε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, μάλλον δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς ε, καλά τους αριθμούς για να δει ποια είναι τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί στην Ελλάδα και πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί. Η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης είναι μια πολύ καλή ιδέα και δεν χρειάζεται να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Ε, θα ήθελα απλώς να πω ότι ε, θα χρειαστεί οπωσδήποτε και η απαραίτητη παροχή μάλλον απαραίτητη τεχνικής αρρωγής έτσι ώστε ε, να απορροφηθούν γρήγορα τα κονδύλια αυτά. Οπωσδήποτε θα πρέπει οι επενδύσεις να αφορούν, να είναι στραμμένα προς το μέλλον, να αφορούν την ανάπτυξη και φυσικά θα πρέπει να μάθουμε όλοι να καταναλώνουμε όχι απαραίτητα περισσότερο αλλά καλύτερα συγχρηματοδότηση είναι μικρό το ποσοστό και είναι απολύτως απαραίτητο οι περιφερειακές και οι εθνικές αρχές να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους και την ορμή τους όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ε, ε, ε, ο κατάλογος των χωρών αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει έξι χώρες μονάχα. Τι θα γίνει εάν στο μέλλον αντιμετωπίσουν δυσχέρειες και άλλες χώρες γιατί βλέπουμε ότι η οικονομική κατάσταση αλλάζει σε πολλές περιπτώσεις. Τι θα γίνει και με ταχύτητα, τι θα γίνει λοιπόν εάν ζητήσουν και άλλες χώρες τη βοήθεια αυτή. Ε, γίνεται λόγος για μη αύξηση ε, των ε, κονδυλίων. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει λιγότερα προγράμματα και επίσης ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί σε αυτήν την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιχαήλ Τρεμόπουλος. Κύριε ε, αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά χαιρετίζω αυτή την ε, απόφαση, αυτό το μέτρο, να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση μέχρι το και το 90% στις, ε, στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, που σήμερα πια είναι σαφές ότι απειλεί ολόκληρη την Ευρωζώνη. Βέβαια, όταν το είχα θέσει εδώ με τη μορφή ερώτηση στον Επίτροπο, τον κύριο Χάν, κάποιοι συνάδελφοι αντέδρασαν. Και τότε ο κύριος Χάν είχε απαντήσει ότι θα το πάμε ε, λίγο παραπάνω, αλλά δεν τολμούσε και αυτός να σκεφτεί το 90%. Συμφωνώ, ε, κύριε συνάδελφοι, ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμο. Δεν μπορεί να είναι ο κανόνας. Άλλωστε δεν συμφέρει. Γιατί δεν συμφέρει. Γιατί δεν αυξάνει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει στις χώρες αυτές, ούτε τα χρήματα παίρνονται από άλλα έτη. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Απλώς μειώνεται η εθνική συμμετοχή. Δηλαδή, το αποτέλεσμα θα είναι να γίνουν λιγότερο, λιγότερα έργα. Αυτό είναι. Το πληρώνει η ίδια η χώρα. Είναι όμως έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και με την ελπίδα ότι θα μπορέσει σύντομα να έχει κάποιο είδους σταθεροποίηση φυσικά και ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν κάνει σοφά η πρόταση αυτή. Να ενισχύσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάποια έργα. Σε μια χώρα όπου η απορρόφηση ήδη είχε πρόβλημα με τα προηγούμενα ποσοστά. Δεν υπήρχαν ίδια κεφάλαια, και λόγω της κρίσης, εγώ θα έλεγα και λόγω μειωμένης ικανότητας. Ναι, είναι σαφές. Έχω μια μακρά θητεία και στην αυτοδιοίκηση, στο δεύτερο βαθμό, και γνωρίζω τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να μας μπρόξει μπροστά. Να βοηθήσουμε, να παρακολουθούμε τα έργα. Να ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν τα μάτια κάποιων. Περάσαμε την έκθεση πέρυσι και ως Επιτροπή και ως Ολομέλεια για την διαφάνεια στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για αυτά που συζητάμε από τα περιφερειακά ταμεία. Η διαφάνεια είναι ξεκαθάρισμα των όρων του παιχνιδιού γιατί ναι, κάποιοι κάναν πάρτι στα προηγούμενα χρόνια. Αυτά πρέπει να κοπούν. Να μπορέσει, να μπορέσει η Ελλάδα και κάθε χώρα που έχει προβλήματα να σέβεται και η εκπροσωπή τη τους όρους του παιχνιδιού. Άρα παρακολούθηση. Άρα υψηλή ποιότητα των έργων που εγκρίνονται. Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Γιατί σήμερα βιώνουμε στην Ελλάδα μία επίθεση στην βιωσιμότητα με πάρα πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα να σας πω να καταλάβετε με τα αυθαίρετα. Υπάρχει εκτεταμένο κτίσιμο αυθαιρέτων στην Ελλάδα, υποτίθεται πληρώνουν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται. Σήμερα χαρίζονται με την ανοχή της Τρόικας δηλαδή της Κομισιόν. Ή γίνονται γενναίες εκπτώσεις για να επιβραβευθεί η παρανομία. Με εντολή της Τρόικας έχει καταργηθεί τα δύο τρίτα του σιδηροδρομικού δικτύου. Γιατί λέει δεν αποδίδουν. Δεν είναι αυτή η λογική πονάει χέρι, κόψει χέρι. Δεν μπορείς να καταστρέφεις τις υποδομές της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Χρειάζεται είπαμε και διαφάνεια και γνώση, σωστή διαχείριση των κονδυλίων και οι χώρες που αδυνατούν ή καθυστερούν υπέρμετρα να μπορέσουν να έχουν αυτή τη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις κακές πλευρές της οικονομίας τους και της νοοτροπίας τους. Χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση, συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, παρακολούθηση της προόδου σχεδιασμού, της απορρόφησης των κονδυλίων, της υλοποίησης των έργων. Ναι, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη για να μπορεί στο τέλος τα λεφτά που δίνεις ή τουλάχιστον κάνεις κόντο για να μπορέσουν να γίνουν κάποια έργα, αυτές οι κινήσεις να μπορέσουν να αποδώσουν. Οι ροές των κονδυλίων και οι επιδόσεις αξιοποίησης είναι ένα τομέα που πρέπει να τον δούμε σοβαρά. Και από χρηματοοικονομική πλευρά είναι σημαντικό να γίνεται λογιστική παρακολούθηση των χρημάτων. Τα έργα να παρακολουθούνται ενώσο υλοποιούνται. Και τέλος να υπάρχει και ενδυνάμεση αξιολόγηση για να μπορέσουμε να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που το λέω τώρα, αλλά πραγματικά δεν θα έχουμε χρόνο αν, αν ε, μιλάμε όλοι πάρα πολύ. Ε, πρώτον, καλωσορίζω, λέει η κυρία Κλέβα, την πρόταση αυτή. Να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη παρατήρηση σχετικά δηλαδή με τις επιπτώσεις αυτής της πρότασης δεν είμαι ακόμα σίγουρη ε, για το τι αντίκτυπο θα έχουν αυτά τα 2,3 δις. Θα ήθελα μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί νομίζω ότι όλοι το σκεφτόμαστε, αλλά ε, δεν το ε, εκφράζουμε. Βεβαίως κανείς εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν είναι κατά της βοήθειας προς τις χώρες οι οποίες χυμάζονται από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ωφέλιμη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως αυτά που είπε και η Πρόεδρος, να μην μακρηγορούμε. Γι' αυτό λέω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την κυρία Μανέσκο και με τον συνάδελφο Όλβριχτ και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Έτσι κι αλλιώς χαίρομαι πάντα όταν συμφωνώ με τόσο σοφούς συναδέλφους. Έχω όμως δύο ερωτήματα. Μια ερώτηση ε, προς το Συμβούλιο και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα και τα όσα μας είπαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, τα πράγματα φαίνουνταν καθυσυχαστικά. αλλά μετά είπε το Συμβούλιο ότι έχει ήδη συνεδριάσει πέντε φορές η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και είναι πολύ κοντά σε αποτέλεσμα. Μα χρειάζεται το Συμβούλιο να συνεδριάζει πέντε φορές την ομάδα εργασίας και παρόλα αυτά μιλάμε στο μέλλον για συμπέρασμα και αποτέλεσμα, Πόσες φορές πρέπει να συνεδριάσει δηλαδή. Μου φαίνεται αντιφαντικό, δεν ξέρω αν είμαι ιδιαίτερα παρανοϊκός, αλλά αν ήταν όλοι οι ομόφωνοι στις πέντε φορές που συνεδρίασε, γιατί συνεδρίασε πέντε φορές η ομάδα εργασίας ε, αρμόδια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω τι συμβαίνει, να έχουμε πληροφόρηση, είμαι υπέρ τη επιταχυμένη διαδικασία, αλλά Για ποιο λόγο παρακαλώ χρειάστηκαν πέντε συνεδριά στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου και μας λέτε ακόμα ότι επίκειται. Πότε δηλαδή. Και για το θέμα της αναδρομικής ισχύω υποτίθεται ότι είστε σύμφωνοι. Άρα τι συζητάτε πέντε φορές στο Συμβούλιο. Και δεύτερη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Βαρόσο κατονόμασε την Ελλάδα αλλά δεν αναφέρθηκε σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Είπε ότι για το Ταμείο Συνοχής θα καταβάλουμε προσπάθεια να κάνουμε και νέες προτάσεις. Και πρόσθεσε ότι για τις προτάσεις αυτές θα γίνουν διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε τίποτα λοιπόν για αυτές τις προτάσεις, έκτοτε για αυτά που ανέφερε το Κοινοβούλιο και ο Σπαρός, οπότε θα καταθέσει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα ήταν ε, απολύτως απαραίτητο, όσο και επίγον, να εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις στα πλαίσια της κρίσης και να τα δούμε όλα συνολικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ βεβαίω να συμφωνήσω με την πρόταση αυτή, αλλά διστακτικά. Γιατί η πρακτική έχει καταδείξει ότι εάν δώσουμε φτηνό χρήμα σε ε, κάποιους, δεν χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά ε, αποτελεσματικά. Επομένως, θα πρέπει η βοήθεια αυτή να έχει πολύ σαφείς κανόνες. Ε, θα πρέπει επίσης να υπάρξουν κανόνες οι οποίοι θα απλουστεύσουν την βοήθεια και ότι σίγουρα η βοήθεια αυτή θα παράγει ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Μήπως θα μπορούσαν να απαντήσουν στα σημεία αυτά όσο γίνεται πιο σύντομα. Κύριε Νίσλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους σας. Λακωνικά θα απαντήσω. Η κυρία Μανέσκου έκανε λόγο ε, για το πακέτο της κρίσης και ποιος θα είναι, είναι ο αντίκτυπος. Έγινε συζήτηση πριν από λίγο καιρό ε, για μία έκθεση με θέμα ακριβώς αυτή την κρίση ε, και ένα ευρύ φάσμα μέτρων οικονομικής και άλλης φύσης. Κυρίως δε έδωσαν κάποιες πληροφορίες σχετικά τι ε, θα μπορούσε να γίνει με τις προκαταβολές καταβολές χρημάτων σε πρώιμο στάδιο. Κύριε Όλμπριχτ, αναφερθήκατε στην πολιτική συνοχή λέγοντας ότι θα μπορούσε ε, να αποτελέσει ένα όχημα ε, το οποίο θα βοηθήσει την έξοδο από την κρίση. Είναι γεγονός αυτό ε, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μία δεύτερη δοκιμασία. Δηλαδή ο στόχος μας είναι τώρα ο επόμενος κανονισμός να περιλαμβάνει τέτοιες διατάξεις ε, που θα επιτρέπουν την ε, ε, υλοποίηση μέτρων υπό εξαιρετικές, υπό συνθήκες. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Θα το δείτε στο προσχέδιο που θα δείτε αύριο. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι μέσω της του μεγαλύτερου ποσοστού ε, χρηματοδότησης ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν ε, λιγότερα έργα. Παρόλα αυτά το σημαντικό για μας, η προτεραιότητα για μας είναι να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση έργων που έχουν ήδη ε, ξεκινήσει έτσι ώστε να ολοκληρωθούν ε, με τα χρήματα αυτά και επίσης ε, να μειωθεί η υποχρέωση χρηματοδότησης από πλευράς των κρατών μελών για τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να αντλήσουν χρήματα από τις ε, εθνικούς ε, πόρους και που πρέπει να δανειστούν κεφάλαια έτσι ώστε να ολοκληρώσουν ε, τα έργα αυτά. τι είναι αυτή η ρήτρα λήξης, η sunset clause. είναι η συμπερίληψη μιας ημερομηνίας που αφορά το τέλος της διαδικασίας και που μπορεί να μην ταυτίζεται με τις ημερομηνίες ελήξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες με το Συμβούλιο. Ε, θα απαντήσω όμως τους κυρίους Αγκουράκη και Τρεμόπουλο. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι τα μέτρα αυτά ε, στην ουσία ε, συμπληρώνουν τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί από ε, ή υπέρ των χωρών που αντιμετωπίζουν ε, κρίση και πριν αναγκαστούμε να τροποποιήσουμε κανονισμούς. Ας πούμε, έχει υπάρξει τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος για την Ελλάδα, του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να υπάρξει μία μετακύληση των δραστηριοτήτων ε, εάν ε, δει κανείς πόσο, με πόσο δραματικό τρόπο έχουν εκτυλιχθεί τα γεγονότα και οι εξελίξεις ε, στην Ελλάδα, ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ανεργία, ξέρουμε πόσο μεγάλη κρίση διανύουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν κάποια μέτρα, κυρίως για τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ε, επαναπρογραμματισμός των δράσεων και επομένως αφού λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα ε, ε, λέμε ότι θα υπάρχει και αυτή η διαφορά στην συγχρηματοδότηση. Σάντσε Σμιτ. Ρωτήσατε τι θα συμβεί εάν και άλλες χώρες ζητήσουν αυτήν την στήριξη. Ο τρόπος διατύπωσης ε, του ε, κανονισμού είναι τέτοιος ε, που αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο χώρες οι οποίες προσφεύγουν στους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να έχουν και αυτού του είδους την στήριξη. Κατά αυτήν την έννοια όμως η συζήτηση για ένα ζήτημα όπως είναι η ρήτρα τέλους, the sunset clause, ε, αποκτά μεγάλη σημασία. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ότι ναι υπάρχει στήριξη αλλά ε, με όριο το 2013. Η κυρία Κλέβα αναφέρθηκε στον αντίκτυπο ε, και στα επιπλέον κονδύλια. Δεν υπάρχει λόγος, δεν γίνεται λόγος για επιπλέον κονδύλια. Μιλάμε για τροποποίηση της ε, πολιτικής και επομένως ε, μια προκαταβολή των χρημάτων και μετά από αυτήν την ε, περίοδο ε, θα υπάρξει ε, οπωσδήποτε μείωση της χρηματοδότησης μέχρι ότου να υπάρξει εξισορρόπηση. Λέμε λοιπόν ότι για κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχει καταβολή εμπροστοβαρής των χρηματοδοτήσεων 15% ας πούμε όσον αφορά τη, την ανταγωνιστικότητα ή λίγο παραπάνω όσον αφορά τη συνοχή και μετά επανερχόμαστε ε, στα κανονικά. Βλέποντας ε, την ε, διαδικασία και βλέποντας την σε προοπτική θα καταλάβετε ότι ενδεχομένως το ποσοστό χρηματοδότησης ίσως να είναι ελαφρά ε, ε, υψηλότερο από το ανώτατο όριο που καταδεικνύεται στους κανονισμούς, αλλά στην ουσία ενδεχομένως η κατάσταση να δυσκολέψει τη στιγμή της εξόδου ε, των χωρών αυτών από τον μηχανισμό. Ο κύριος Ντόιτς αναφέρθηκε στις δηλώσεις Μπαρόσο Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει τελειώσει η κρίση. Και προσπαθούμε να δούμε όλες τις δυνατότητες που μας ανοίγονται ε, για το μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να παράσχουμε τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα, θα... θα είναι απαραίτητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η κυρία Μανέσκου νομίζω ότι δεν κατάλαβε την απάντησή σας ε, ή δεν είναι ικανοποιημένη. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομη θα είμαι. Θα ήθελα να θυμίσω στον κύριο Νίσλερ, αν μου επιτρέπει, τη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν έμεινα ικανοποιημένη από την ανάλυση σας, διότι βασίζεται μόνο σε στοιχεία αριθμητικά που σας δίνουν κυβερνήσεις. Και σας είχα ρωτήσει ήδη από τότε. Πιστεύουμε και βασιζόμαστε μόνο στα στοιχεία των κυβερνήσεων. Τότε μας είπε ο κύριος Νίσλερ ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτά έχουμε μόνο στοιχεία λάβει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γελιόμαστε ή να εθελοτυφλούμε γιατί μπορούμε να οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα διδασκόμαστε από την εμπειρία ότι αυτά που μια φορά δηλώνουν ως στοιχεία κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα. Και εγώ περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια νυφάλια όσο και πραγματική αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε επίσης πολύ σύντομα. Δύσκολη ερώτηση, κυρία Μανέσκο, όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια πολιτική που είναι υποκοινή διαχείριση και βασίζεται σε σχέσεις που είναι σχέσεις εμπιστοσύνης κανονικά και διαφάνειας ως προς τα στοιχεία που μας δίδουν. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν απαιτήσει αναφοράς ε, από πλευρά κρατών μελών που είναι υποχρεωμένα να διαβεβάζουν πληροφορίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια εμεί να εκτιμούμε την κατάσταση στο εκάστοτε κράτο μέλο. Δηλαδή, όταν πρόκειται για την ε, εκτίμηση ε, των μελλοντικών εξελίξεων, βασιζόμαστε στα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη με τις εκθέσεις υλοποίηση και τις αναφορές. Και φαντάζομαι ότι το κατανοείτε αυτό. Τελευταία παρατήρηση. Έχουμε συνολική ευθύνη να αξιολογούμε και να υπολογίζουμε τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής. Όπως γνωρίζετε με περιοδικό τρόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αυτόματα ή γενικά, συνολικά. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ως προς το γιατί πέντε συνέδριο του Συμβουλίου τώρα. Η απάντηση είναι απλή. Εξετάσαμε επισταμένως όλες τις λεπτομέρειες σε τουλάχιστον τέσσερις τομείς που μπορώ να αναφέρω. Ο πρώτος είναι οι επιπτώσεις επί του προπολογισμού συζήτησαμε συγκεκριμένα τον αναδρομικό χαρακτήρα και την ρήτρα λήξης. Ο τομέας είναι η εμπλοκή της Κομισιόν στην διαδικασία, γιατί η Κομισιόν έχει προτείνει την αυτόματη ενεργοποίηση του μηχανισμού, το συζήτησαμε και αυτό. Ένας άλλος τομέας, ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε στην ομάδα του Συμβουλίου, αφορούσε την νομική μεθόδευση ώστε τα κονδύλια αυτά να προαγάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και τέταρτος, τέταρτη θεματική ενότητα, να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά όντως χρειάζονται στην εκάστοτε χώρα. Αυτά τα θέματα μας απασχόλησαν στις πέντε συνόδους του Συμβουλίου. Κύριε Χόμπλερ, ευχαριστώ πολύ όσοι εισηγήτρια να πω δύο κουβέντε. Μετά από τις συναντήσεις με το Συμβουλίο και την Κομισιόν και μετά από την πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές χθες, προετοιμάσαμε τροπολογίες επί τεσσάρων θεματικών ενωτήτων. Ε, ο προαιρετικός, ο χαρακτήρας με την ρήτρα λήξης μας απασχολεί να δούμε ποια είναι η καλύτερη επιλογή γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια στο τραπέζι. Δεν τα συζητήσαμε εδώ αλλά πρέπει να δούμε τελικά τι επιπτώσεις έχουν αυτοί οι δύο όροι στο ύψος των κονδυλίων και στον χρονισμό της μεταφοράς τους. Μετά ο αυτοματισμός, εγώ γενικώ είμαι υπέρ, ε, όχι πλήρους αυτοματισμού, αλλά υπέρ μιας πολύ ευέλικτης διαδικασίας, μιας απλής διαδικασίας, χωρίς γραφειοκρατία δηλαδή για την ενεργοποίηση του μηχανισμού, όχι στα γραφειοκρατικά εμπόδια, κάτι το οποίο απασχολεί δηλαδή ελάχιστα την Κομισιόν. Ως προς το τρίτο, Και εδώ έχουμε διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα αναφοράς, υποβολή εκθέσεων κλπ. Γι' αυτό λέω για άλλη μια φορά να προσφύγουμε στον υφιστάμενο μηχανισμό παρακολούθησης. Ε, Τρει ήταν μίσο, μάλιστα δεν ήταν τέσσερι, λάθο δικό μου λέει κύριε Χούμπνερ. Πολύ ωραία. Πρόθεσμη υποβολή τροπολογιών 14 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου και προς τους Κιώδης να πω ότι μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, φέρνουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρόνο, αλλά θα καθυστερήσουμε το μέθε επόμενο κατά 10-15 λεπτά για να αφιερώσουμε τουλάχιστον μισή ώρα στο επόμενο. Και πάλι η τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά την χρηματοοικονομική τεχνική, το financial engineering, ουσιαστικά πρόκειται για τις ε, επιστρεπτές ενισχύσεις. Για να μην επαναλάβω τα γνωστά, ε, ο κύριος Νίσλερ πιστεύω θα είναι καλύτερο να μας μιλήσει ο ίδιος. Ρούντουλφ. εδώ πρόκειται για μια τελείως διαφορετική πρόταση. Η λύση που προτείνουμε εδώ είναι τεχνικής φύσεως βασίζεται σε έβριμα του Ελληνικού συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο κράτη-μέλη, τα οποία απολαύουν επαναλαμβανμένων μέτρων υποστήριξης, προβαίνουν σε ενισχύσεις, οι οποίες οικονομικής απόψεως δεν συνάδουν με το άρθρο 44, όσον αφορά δηλαδή τα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής και όσον αφορά την διάρθρωση των ταμείων τα οποία επενδύουν απευθείας έργα. Αυτές οι δράσεις και τα συναφή έργα τελούν υποαίρεση, υπάρχουν αμφιβολίες δηλαδή όσον αφορά την χρηματοδότησή τους, κατά πόσο χρηματοδοτούνται νομίμως. Η Κομισιόν λοιπόν μαζί με τα κρατημέλη διερεύνησαν την κατάσταση. Εξετάσαμε δηλαδή τα συγκεκριμένα κρατημέλη για να δούμε πώς χειρίζονται τα κρατημέλη αυτά τα έργα και βεβαίως και εμείς οι νομικοί μας κατήσαμε και εξετάσαμε τι καλύπτει ο κανονισμός και τι δεν καλύπτει. Τι είναι επιλέξιμο και τι όχι. Διεπιστώσαμε, καταλήξαμε στο ότι όντως υπάρχουν αρκετές δράσεις που υλοποιούν τα κρατημέλη, τα οποία είναι συνέχεια δράσεων της περίοδου πριν το 2007. Κάποιοι χρονολογούνται ήδη από το 1994. Αυτές οι δράσεις ήταν πλήρως επιλέξιμες με βάση τον προηγούμενο κανονισμό και εκεί υπάρχει και η σχετική νομική βάση. Εκεί είμαστε εντάξει. Εδώ μιλώ αποκλειστικά για τα παλιά, αν θέλετε, κρατημέλη, τα οποία καλή την πίστη και βάση του κανονισμού χρηματοδότησαν αυτές τις δράσεις που αν θέλετε δεν απαγορεύονται ρητός από τον κανονισμό. Και έτσι ουσιαστικά μετακυλήθηκε αυτή η πρακτική στο τωρινό πλαίσιο. Επίσης οι νομικοί μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα παραθυράκι, ένα νομικό κενό στον κανονισμό που δεν εξής ανεξαρτήτως του ότι δεν απαγορεύονται αυτές οι δράσεις, δεν υπάρχουν από την άλλη πλευρά διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τη χρήση ακριβώς επιστρεφωμένων ποσών για τις κυλιόμενες αυτές δράσεις. Οπότε, προσπαθήσαμε να προβούμε σε μια διορθωρική διορθωτική δράση μέσω αυτής της τροπολογίας για να εξασφαλίσουμε στα κράτη-μέλη τη νομική ασφάλεια η οποία θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την υλοποίηση αυτών των δράσεων με τρόπο μη αμφισβητήσιμο και σύμφωνο με τις καλές πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει σε προηγούμενες περιόδους. Και τούτο γιατί σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις προσπάθειες να αξιοποιηθούν τα κοινωτικά κονδύλια με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και οι ενλογοδράσεις είναι δράσεις που έχουν τέτοιο αποτέλεσμα. Η πρότασή μας λοιπόν αφορά στην διόρθωση αυτού του νομικού κενού. Επιπλέον, αποφασίσαμε στο ίδιο πλαίσιο να προβούμε σε μερικές διευκρινήσεις του κανονισμού. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε σημεία τα οποία διέπουν τις σχέσεις μας με τα κρατημέλη ε, όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα κρατημέλη σε θέματα χρηματοοικονομικής τεχνικής, για παράδειγμα. Έτσι επενεύουμε εκεί που χρειαζόταν στον κανονισμό με τροπολογίες. Και επιπλέον παραφέρουμε συγκεκριμένε διατάξεις τις οποίες συνομολογήσαμε με τα κράτη-μέλη επιθελοντικής βάσεως. Και τούτο γιατί, για παράδειγμα, η υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών τεχνικών. Είναι θέμα το πώς χρησιμοποιούνται τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ξέρετε, πολλές φορές δεν, υπήρχε υποχρέωση, δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και εκεί συνειδητοποίησαμε κάποια στιγμή ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για να μπορέσουμε να προβούμε ακριβώς την παρακολούθηση της χρήση αυτών των μέσων. Και αυτό προέκυψε κάποια στιγμή στις επαφές που είχαμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Προτείνουμε λοιπόν να θεσπίσουμε μια, ένα εθελοντικό μηχανισμό υποβολής εκθέσεων ο οποίος τώρα γίνεται υποχρεωτικός όμως για τα κράτη-μέλη. Επίσης, για να βοηθήσουμε στην κατάρτιση της ετήσιας δήλωσης αξιοπιστίας προσθέσαμε υποχρεώσει που έχουν σχέση ακριβώ με αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και τι προκαταβολές στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και τούτο με στόχο και πάλι ο αρμόδιος χειριστής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, να μπορεί να έχει σαφή εικόνα των οριασμών. Πιο συγκεκριμένα, θέλουμε να είναι σαφής η διάκριση των προκαταβλών, για παράδειγμα, από άλλες δαπάνες. Πρόκειται για πληροφορίες, αν θέλετε, που δεν είχαμε παλιά στη διάθεσή μας, με τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονταν οι εκθέσεις στο πλαίσιο πάνω της διαδικασίας πληρωμών. Επίσης, προτείναμε επιπλέον προτείναμε, όπως ε, έλεγα, οι πληρωμές αυτές μέσω χρηματοοικονομικών τεχνικών είναι σαφές εάν πηγαίνουν σε ενδιαμέσους ή στους τελικούς δικαιούχους, στους τελικούς μάλλον αποδέκτες. Προσθέτουμε λοιπόν διάταξη που προβλέπει ότι οι πληρωμές δεν μπορούν να κατακατούνται πάνω από δύο χρόνια σε τέτοιου είδου ταμεία ενδιαμέσους. Υποβάλλουμε αυτή την πρόταση εν γνώση μας ότι αυτό θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί πρακτικά στη φάση αυτή, ε, εφόσον δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτές οι δράσεις. Και δεδομένου ότι ήδη έχουν προκριθεί συγκεκριμένες συμβατικές ε, ε, συμφωνίες μεταξύ των αρχών και των ενδιαμέσων αυτών αρχών ταμείων. Και αυτό το συζήτησαμε στο Συμβούλιο μαζί με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, η οποία είπε ότι αυτή η διάταξη μπορεί από νομικής απόψεως να μας δημιουργήσει μάλλον προβλήματα. Εν τούτης, όσον αφορά αυτήν την περίοδο των δύο ετών, πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ενώ ότι τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν το βάσιμο αυτού του αιτήματο, της υποχρέωση δηλαδή, και συμφώνησαν στις μελλοντικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές τεχνικές αυτό το κριτήριο να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί. Εμείς ακούσαμε τα κράτη-μέλη και, τους, και την νομική υπηρεσία και με βάση αυτά η Κομισιόν απέσυρε την αρχική της πρόταση παρά το γεγονός ότι την κρατάμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο γιατί θεωρούμε ότι έχει λόγο ύπαρξης. Σκοπεύουμε η Κομισιόν να προβεί σε επίσημη δήλωση με την οποία θα διασφαλίζεται ότι το σημείο αυτό θα ασφαλωθεί στο επόμενο πακέτο για τα διαθροτικά ταμεία. Όταν έρθει η ώρα δηλαδή της νέας από τη διαδικασία στο Συμβούλιο μπορείτε να κρατήσετε ότι η συζήτηση ήταν εξαιρετικά επικοδομητική. Επαναδιατυπώσαμε ορισμένα τεχνικά σημεία του κειμένου για να γίνει πιο αυτοσυνεπές, ώστε να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις σωστά. Στην αυτή κατηγορία λοιπόν των επιστρεπτών ενισχύσεων. Επίσης, τις διατάξεις χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις δηλώσεις δαπανών τις αναδιατάξαμε έτσι ώστε από πλευρά διοικητικών διαδικασιών να είναι πιο ευανάγνωστη κατάσταση, πιο σαφής. Ξεχωρίσαμε λοιπόν αυτά τα δύο τμήματα. Ε, η Κομισιόν επίσης δέχθηκε. Αν το κρατός μέλος είναι πλέον υποχρεωμένο να υποβάλει ετήσια έκθεση για την πρόοδο υλοποίησης των χρηματοοικονομικών εργαλείων, σε αυτήν την περίπτωση η Κομισιόν θα υφετεί αυτά τα στοιχεία και αυτό θα αποτελεί και την έκθεση της Κομισιόν. Έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς την πρόοδο, την υλοποίηση του μέτρου. Κύριε Ζελέντη, είδα την έκθεσή σας και τις προτάσεις σας και τις τροπολογίες και θα έλεγα εκ πρώτη όψη ότι οι περισσότερε τροπολογίε ε, συνάδουν με τι ανάγκε του θέματο και μπορούν να ενσωματωθούν κάλλιστα στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε επικοδομητικά πάνω στο κείμενο, πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ από την πλευρά μου είμαι στην διαθεσή σας για να σας ενημερώσω ή για να συμμετάσχω και σε οποιαδήποτε σύσκεψη. Το κείμενό σας πάντως ε, μου φαίνεται εξαιρετικό και μπορούμε να προχωρήσουμε πάνω στη βάση του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόιτα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την τροποποίηση την έχουμε συζητήσει ήδη. Το είπε και η κυρία Χιούπνερ προηγουμένως. Ως εισηγήτρια ότι οι σκιώδεις εισηγητές το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Και εγώ είχα καταλάβει ότι συμφωνήσαμε όλοι να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη αυτή την τεχνική προσαρμογή, ακόμα και αν υπάρχουν αντιστάσεις ε, γιατί είναι μια ασφάλεια για εκείνους που κάνουν αυτές τις ανανεώσιμες πιστώσεις, τα revolving credit Fund. Ε, και ε, θα ήθελα να πω κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να γίνει με τέτοιο τρόπο η προσαρμογή για να μην παρεμποδίζεται το εργαλείο αυτό καθ' αυτό το μέσο. Υπάρχουν από χώρα σε χώρα διαφορές. Μερικοί το θεωρούν βουνό, τεράστιο πρόβλημα ε, πού θα γίνουν εκταμιεύσεις, πού θα πηγαίνουν τα κονδύλια. Αυτό δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε πολύ συγκεκριμένα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Γρήγορα να προχωρήσει μεν η προσπάθεια, αλλά από την άλλη θέλω να διαφυλαχθούν και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ε, και να μην τρέχουμε συνέχεια στο ελεκτικό συνέδριο ε, για να λύνουμε τις διαφορές μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό θα ήταν εις βάρος αυτής της ιδέας των ανανεώσιμων πιστώσεων. Από τη μια κατάλαβα εγώ λοιπόν ότι αυτή τη διετία ε, που το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, τώρα δεν γίνεται να το επιβάλλει γιατί δεν της επιτρέπεται. Μετά μας είπατε ο τρόπος που θα γίνονται οι αναφορές και οι εκθέσεις. Ε, συνάδει ε, με τη νέα διαδικασία. Η κυρία Χιούμπνερ έχει κάνει αλλαγές, έχει απλοποιήσει πάρα πολύ. Αυτό σας ικανοποιεί, είναι αρκετό ή ε, υπάρχουν και άλλα θέματα σημαντικά έτσι ώστε ε, αυτή η ιστορία με το Ελεκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου να λειτουργήσει. Και θέλω να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την τροποποίηση που προτείνεται με ΑΙ συμφωνεί, μπορεί να μας πει ότι υπαρκούν οι πληροφορίες που έχει. Περνάει από το Συμβούλιο και είναι εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και εμένα προσωπικά είναι το εξής. Πρώτον, θα πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουν τελικά τα κονδύλια σε ποιο φορέα, εν πάση περιπτώσει, καταλήγουν τα ευρωπαϊκά χρήματα που είναι δημόσια οι και επίσης πώς δαπανάτε αυτό το χρήμα και ποιο είναι το ποσοστό που αναλογεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω την έκθεση διαφάνειας που έκανε το Κοινοβούλιο σχετικά. Για μας είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να κινηθούμε. Βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα φουσκώσουμε και τη γραφειοκρατία διότι ε, πρόκειται για μικρά έργα, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, σε αυτή τη τεχνική, ε, τη χρηματοπιστωτική. Και είναι κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω καθόλου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα του άρθρου 44α δεν ζήτησε να εφαρμόζονται διάφορες διατάξεις που αφορούν και το άρθρο 57 του ισχύοντος κανονισμού διότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τα έργα που ήδη χρηματοδοτούνται από το μέσο αυτό. Εμείς ε, θέλουμε να απαλληφθεί αυτή η διάταξη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει. Ο κύριος Τρεμόπουλος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά και να εστιάσω στο ζήτημα των έγκαιρων αποταμιεύσεων και των ρυθμών απορρόφησης από τα κράτη-μέλη που επιδιώκουν αλλά αδυνατούν να χειριστούν με επιτυχία είτε αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στη διαδικασία. Πολλές φορές προχωράει ο σχεδιασμός, Παρουσιάζονται όμως μεγάλες καθυστερήσεις σε αυτό το επίπεδο των μορφών των επιστρεπτέων επιδοτήσεων. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες μπορούν να υπάρξουν. Είδαμε ικανοποίηση ότι υπάρχει πρόβλεψη για νομική υποχρέωση ή χρηματοδοτική συνδρομή που καταβάλλεται από την διαχειριστική αρχή για τη σύσταση ή συμβολή στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιείται για επιλέξιμες δαπάνες μέσα στο χρονικό πλαίσιο δύο ετών από την πληρωμή στο Ταμείο. Αν δεν επιτευχθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα αφαιρούνται τα ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί. Αυτό είναι ένα βήμα άμεσο, σημαντικό. Πρέπει όμως προηγουμένως να εξασφαλίσουμε και άλλες πιο ήπιες μορφές παρεμβάσεων. Για παράδειγμα διαφάνεια που ανέφερε και η κυρία Σρέντερ και ανέφερα και εγώ πριν. Θα πρέπει να δίδονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία από τις αξιολογήσεις που ούτω ή άλλως στέλνουν στην Κομισιόν τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές τους αρχές για την πρόοδο των εργασιών. Θα μπορούσε να γίνεται τακτική και δυναμική αναφορά προόδου ή έστω με ενδιάμεσες εκθέσεις που θα δημοσιεύονται και θα παρουσιάζονται όπου είναι απαραίτητο. Αυτό θα είναι ένα άμεσα καθοριστικό, καθολικό σύστημα παρακολούθησης χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη γραφειοκρατία αφού τα στοιχεία ούτως ή άλλως τα παίρνετε από τις χώρες και θα γίνονταν και γνωστό ποιοι βρίσκονται σε καλό δρόμο, ποιοι υστερούν κλπ. Χρειαζόμαστε δηλαδή βήματα και προτάσεις υλοποιήσιμες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλέβα. Νομίζω ότι θα είστε, ελπίζω να είστε πάλι σύντομοι όπως και την προηγούμενη φορά. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την πρόταση αυτή, κυρίως δε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απλούστευση, την ελάφρυνση του γραφειοκρατικού άχθου, του διοικητικού μάλλον άχθους. Πιστεύω ότι η χρήση αυτού του μηχανισμού θα πρέπει να ενταχθεί σωστά στα υπάρχοντα προγράμματα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ερώτημα των, στο ζήτημα των δύο ετών που αναφέρθηκε ήδη, απλώς αυτό που σας ρώτησα. Νομίζω θα ξαναρχίσουμε πάλι με την Επιτροπή και μετά με το Συμβούλιο. Πρώτα η Επιτροπή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το ζήτημα των δύο χρόνων. Όταν το προτείναμε, ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο σημείο. Ε, ε, τέθη στην συζήτηση που είχαμε με το ελεγκτικό συνέδριο βάσει των ευρημάτων και ξέραμε ότι τα χρήματα θα πρέπει να προωθούνται με ταχύτερο ρυθμό στα πλαίσια των ε, εργαλείων, χρημα... των εργαλείων χρηματοδότησης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια πρώτη προσπάθεια εγκαθίδρυσης τέτοιων εργαλείων, κυρίως σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τέτοια εμπειρία. Έτσι, και αυτό το, το γεγονός δηλαδή την πρώτη φορά ίσως εξηγεί κάποιες καθυστερήσεις. Συνολικά πάντως προέκυψε ότι είναι ένα ζήτημα και ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος ε, που θα ταυτίζεται με την διαθεσιμότητα των χρημάτων. Είχαμε την εντύπωση ότι θα προέκυπτε και τελικά όντως φαίνεται και στη ζήτηση που είχαμε με τα κράτη-μέλη είναι ότι το τελευταίο ε, ότι η αργοπορημένη εφαρμογή της ε, πρότασης ε, ε, κινδυνεύει να θέσει ε, εν κινδύνο κάποια προγράμματα, ειδικά όταν ε, έχουν ήδη αναλυφθεί υποχρεώσεις, όταν έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια έργα, έστω και αν έχουμε πολύ καλές προθέσεις όσον αφορά την πειθαρχία, πραγματικά θα πρέπει να αποφύγουμε οτιδήποτε θα δημιουργήσει ανομαλία στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Απ' την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι η νομική ασφάλεια και οι ε, νόμιμες πούμε ε, προσδοκίες των ενδιαφερομένων είναι κάτι που μας αφορά και δεν θέλουμε η κατάσταση να ε, αλλάξει. Όμως είναι γεγονός ότι στο, στον επόμενο κανονισμό ε, θα υπάρχουν τέτοιου είδους ε, πρόνοιες ε, σχετικά με την επιθαρχία τη στιγμή που θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Η κυρία Σρέτερα αναφέρθηκε στην απλούστευση της, του τρόπου αναφοράς. Όντως πρέπει να απλουστευθεί λίγο η πρόταση μέχρι τώρα. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί σε αυτό το σκέλος όταν δίνεται επιπλέον πληροφόρηση μέσα, αυτό γίνεται στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ε, πληρωμής. Επομένως, η Κομισιόν θα είναι σε θέση να ε, ζητήσει και να πάρει πληροφορίες όταν αυτές είναι απαραίτητες, έτσι ώστε η λογιστική εργασία να γίνει σωστά σε περίπτωση που η καταβολή θεωρηθεί προκαταβολή και πρώιμη καταβολή, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να έχουμε αυτή τη διαδικασία αναφοράς. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει απλούστευση και το θέμα του χρονοδιαγράμματος δεν παίζει πλέον ρόλο. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να απλουστεύσουμε το συνολικό σύστημα ε, αναφοράς ε, και έτσι ώστε να κρατήσουμε τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές αναφοράς. Ε, αυτό θα γίνεται λοιπόν στο μέσο του έτους και η Κομισιόν δέχτηκε ότι βάσει αυτών των αναφορών μάλλον ότι ε, αυτές οι αναφορές θα γίνονται ε, μέχρι τον Οκτώβριο και ε, βάσει των πληροφοριών που θα έχουμε από τα κράτη-μέλη, βάσει αυτών των πληροφοριών θα προχωρούμε σε μία ενδιάμεση ενημέρωση. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη πάρει από τα κράτη-μέλη βάσει αυτής της εθελοντικής διαδικασίας αναφοράς. και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στους ερχόμενους μήνες θα έχουμε ε, και στη διάθεσή μας ε, θα δημοσιεύσουμε και την πρώτη τέτοια ε, έκθεση. Η κυρία Σρέτερ, βάσει του εθελοντικού συστήματος αναφοράς, η κυρία Σρέτερ έκανε και μια άλλη ερώτηση σχετικά με την μη εφαρμογή του άρθρου 39 56 και 57 και εσείς αναφερθήκατε στο 57 για τα οικονομικά εργαλεία. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι πρόνοιες που βάζουμε στον κανονισμό, τις βάζουμε ε, για λόγους ε, διασάφησης. Γιατί τους γνωρίζουν ήδη τα κράτη-μέλη. Ε, τα, αυτά τα τρία άρθρα αφορούν τα μεγάλα, τα κύρια προγράμματα, τα προγράμματα τα οποία δημιουργούν θέσεις εργασίας. Όταν κανείς φέρει στο νου του τα ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή των άρθρων ε, ε, ένα, ένα ταμείο δεν είναι μεγάλο πρόγραμμα, δεν μπορεί να συγκριθεί, αν θέλετε, με κάποιο δάνειο που δίνεται σε μια επιχείρηση. Ε, και που ενδεχομένως μπορεί να καλύψει και το κόστος ας πούμε ε, της μετεγκατάστασης ε, της επιχείρησης αυτής σε μια άλλη χώρα. Εδώ η λογική είναι διαφορετική και επομένως αυτού του είδους οι δεν έχουν έννοια νομίζω ότι απήντησα και ήδη την ερώτηση του κύριου Τρεμόπουλου σχετικά ε, με, την, ε, τον τρόπο ε, αναφοράς. Σας είπα ότι εμείς βασιζόμαστε σε αναφορά που με τα κράτη-μέλη. Πριν να δώσω ένα λεπτό στο Συμβούλιο, να πω ότι αν στο μέλλον αποφασίσουμε υπέρ αυτής της περίοδου των διετών, τότε πρέπει να έχουμε και κάποια ιδέα του τι θα κάνουμε με τα χρήματα αυτά, εάν μετά τα δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν δαπανηθεί. Λοιπόν, δεν σας δίνω το λόγο. Ένα λεπτό μόνο στο Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε η Κομισιόν. Απλώς επιβεβαιώνω τα όσα είπε ο Ρούντελφ Νίσλα Και προσθέτω ότι στο σχέδιο εκθεσή σα. και στις τροπολογίες βλέπω πράγματα τα οποία συμφωνούν να ε, συνάδουν με τη δική μας συλλογιστική με τη θέση γενικά που, έχουμε, που έχει δημορφωθεί στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα συζητήσεως προθεσμία υποβολής τροπολογιών 14 Οκτωβρίου από την Κομισιόν και το Συμβούλιο κρατώ την υπόσχεση ότι αν χρειαστεί θα συνεδριάσουμε επί του θέματος. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Οπότε προχωρούμε αν και μας μένει λιγότερος χρόνος για το ενδεχομένω σημαντικότερο τη σημαντικότερη μελέτη που έχουμε κάνει όσον αφορά την μελλοντική μας πολιτική. Καλωσορίζω τον δόκτρα Μπάχτλα και τον δόκτρα Μέντες. Είναι, είναι εδώ. Ο κ. Μέντες ίσως όχι. Ο λόγος στον, κύριο, στον δόκτρα Μπάχτλα. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon, members Um, Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Το ο Τζον Μπάχτλα, έστερα ε, μου είναι ο κύριος Μέντες, συναδελφός μου, και οι δύο από το Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Η κυρία Βούσλη, ε, και διάφοροι άλλοι εμπειρογνώμονε μα ε, βοήθησαν πάρα πολύ. Όσον αφορά την ε, παρουσίασή μου, να σου πω ότι θα μιλήσω κυρίω για το μέλλον τη πολιτική συνοχή στο πλαίσιο τη γενικότερη αρχιτεκτονική της πολιτικής μας και τη πολιτική για τον ε, προπολογισμό. Ο Δ. Μέντες στη συνέχεια θα αναφερθεί στο περιεχόμενο αυτής της πολιτικής. Πρόκειται για μελέτη με πολλέ λεπτομέρειε, με πολλέ πληροφορίε. Θα σα μιλήσω επιγραμματικά λοιπόν για τα κύρια ζητήματα από τα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση για το μέλλον τη πολιτική μα. Είναι και τα θέματα τα οποία θα μα προσφολήσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Η δομή είναι ανάλυση πολιτικής. Σταθμίζουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών λύσεων για να κατανοήσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. Αναλύσαμε συστηματικά ακαδημικά συγγράμματα, νομοθετικά κείμενα, μελετήσαμε μοντέλα δαπανών και προπολογισμού, λάβαμε υπόψη μας τους βασικούς περιορισμούς, Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι χρειάστηκε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μα τον Αύγουστο, πριν αρχίσουν να υποβάλλονται δηλαδή τα σχέδια του σχετικού κανονισμού. Βλέπετε εδώ τις βασικές, τα βασικά κεφάλαια της μελέτης, αρχιτεκτονική πολιτική, η εδαφική διάσταση, η στρατηγική συνοχή, οι λεγόμενες αιρεσιμότητε, τα σύνολα προποθέσεων παρακολούθηση, αξιολόγηση, προσθεμένη αξία κ.ο.κ. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Οράματα και εναλλακτικές πολιτικές». Πριν συζητήσουμε το δεύτερο, να τονίσω ως όραμα ότι εγώ με δίστανται όσον αφορά τον σκοπό αυτής της πολιτικής. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πολιτική συνοχή είναι η αναδιανομή των κονδυλίων του προπολογισμού. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι στόχος της πολιτικής είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εδαφικής πολιτικής συνοχής με σκοπό την ανάπτυξη. Μία άλλη διαφωνία αφορά τον ρόλο της πολιτικής εν ώψη της Ευρώπης του 2020. Και εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις που προέρχονται από διστάμενα οράματα όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ της τομεακής και της εδαφικής προσέγγισης, όπως και την το, το δίλημα μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. Όλα αυτά θίγονται στην έκθεση. Θα δείτε εδώ τις διαφορετικές αναλυτικές μας προσεγγίσεις ως προς το πώς πρέπει να εξελιχθεί η πολιτική συνοχή. Επάνω αριστερά, για παράδειγμα, βλέπετε το λεγόμενο δαφικό, την εδαφική συμβατική προσέγγιση Εκεί η πολιτική συνοχή ε, γίνεται αντιληπτή ω ένα εργαλείο υλοποίηση τη πολιτική μα για το 2020. Κάτω αριστερά βλέπετε αντιθέτως μια εδαφική αλλά πιο ριζοσπαστική προσέγγιση με μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών αρχών όπου τα συμφέροντά τους λαμβάνονται υπόψη με πιο έντονο τρόπο σε ενδιαστολή με την κεντρική διαχείριση. Δεξιά βλέπετε την αντίθεση, τους αντίποδες της εδαφικής προσέγγισης. Είναι η τομεακή προσέγγιση. Έχουμε τον τομεακό λειτουργισμό. Είναι μια κεντρική προσέγγιση από το κέντρο προς τα κάτω, από την κορυφή προς τα κάτω, ανεξαρτήτως της εδαφικής συνιστώσας η οποία χαρακτηρίζει για παράδειγμα την προσέγγιση της Παγκόσμια Τράπεζας, τουλάχιστον τη χαρακτηρίζει ως πριν λίγα χρόνια. Και τέλος έχουμε μια ήπια συντονιστική προσέγγιση, τομείς αλλά και συντονισμό από τη βάση προ τα πάνω σε κάποιο βαθμό. Αυτά είναι τα πολύ γενικά. Είναι διαφορετικέ αντιλήψει και διαφορετικέ προσεγγίσει ω προ το τι πρέπει να είναι η πολιτική συνοχή, τι πρέπει να κάνει και πώ σχετίζεται με την Ευρώπη 2020. Ας έρθουμε τώρα στην αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Ένας από τους στόχους της μελέτης μας είναι να διευκολύνει τον διάλογο σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά για παράδειγμα την επιλεξιμότητα και την χρημεροδότηση των περιφερειών. Στη φάση αυτή είναι δύσκολο να πούμε οτιδήποτε γιατί δεν έχουμε τι πληροφορίε ή τι ε, υποθέσει εργασία στην οποία θα κινηθεί η τις υποθεσεις εργασια απο τον οποιο Όμως, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, κυρίως από το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2020, βλέπουμε ότι η αρχιτεκτονική και ο χάρτη εν τέλει τη ε, πολιτικής συνοχής θα έχουν περίπου αυτήν την μορφή. Φαίνεται καταρχήν ότι ο ορισμός των περιφερειών σύγκλησης, δεν θα τροποποιηθεί. εκτός αν ληφθεί υπόψη στην Ευρώπη των 27 αντί των 25. Δεύτερον, οι τρέχουσες ρυθμίσεις για τις ε, περιφερειές μετάβασης θα καταργηθούν. Θα δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία περιφερειών σε μετάβαση, όπου θα είναι μέσα η περιοχές σύγκληση, η περιφέρειες σύγκλησης που ήταν εκεί ως το 2013, όμως εκεί το κατόφλι είναι στο 75% πλέον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κατά κεφαλήν φυσικά, και θα έχουμε εκεί και άλλες περιφέρειες και άλλες περιφέρειες των οποίων το εισόδημα είναι μεταξύ του 75% και του 90% του μέσου κοινοτικού όρου κατά κεφαλήν. Για το Ταμείο Συνοχής το κριτήριο θα είναι το ίδιο μόνο που θα βασιστεί στο μέσο όρο της Ευρώπης των 27 και όχι βεβαίως των 25. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Για το Ταμείο Συνοχής, καταρχήν, φαίνεται ότι βάσει των στοιχείων 2008-2010, 13 κράτη-μέλη είναι επιλέξιμα, για τη συνοχή παραλαμβάνω, τα 12 μέλη χωρίς την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Εν ώψη της νέας διαπραγμάτευσης, η Κύπρος μάλλον θα υποφεληθεί από αυτέ τι μεταβατικές διατάξει. Τώρα όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και την επιλεξιμότητα, τα πράγματα εδώ είναι πιο πολύπλοκα, διότι δεν διαθέτουμε τα τελευταία στοιχεία για το περιφερειακό ΑΕΠ, για το ΑΕΠ κατά περιφέρεια, Έχουμε τα παλιά στοιχεία μέχρι το 2009. Από εκεί πέρα έχουμε μόνο προβολές. Εδώ κεντρική ιδέα είναι ότι θα μειωθούν οι χώρες σύγκλησης Και αυτό θα πειράσει σημαντικά το χάρτη τη επιλεξιμότητα, όπω βλέπετε και εδώ, εξαιτία και τη νέα κατηγορία των περιοχών μετάβαση. Περιοχών με συγχωρείτε μετάβαση. Είχαμε τι περιοχέ που ονομάζαμε λιγότερο ανεπτυγμένες, η κάλυψή του. από 32% του πληθυσμού της ΕΕ θα πέσει στο 24%. Και από 18 κρατημέρια θα πέσουμε στα 16%. Η Γερμανία και η Μάλτα δεν είναι πλέον σε κανένα βαθμό κράτη σύγκλησης. Έτσι Έχουμε αλλαγή σε πολλέ χώρε. 8 δεν θα υποστούν καμία αλλαγή. Τώρα οι σε μετάβαση, οι σε μετάβαση. Εδώ θα αλλάξει ο χάρτη σημαντικά. Πρώτον, όταν λέμε χώρε περιφέρειε μάλλον μετάβαση, Μιλάμε για περιοχές που είναι τώρα στη σύγκληση και οι οποίες όμως δεν αναμένεται να είναι στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια πληθυσμό στην Ευρώπη των 27. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του πληθυσμού είναι στη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία. Η κατηγορία αυτή είναι επίση σημαντική για την Σλοβενία και την Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία θα συμπεριλάβει και άλλες περιφέρειες με ΑΕΠ μεταξύ 75% όπως είπα και 90% του κοινοτικού κατακεφαλήν μεσού όρου. 44 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν, 9% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης των 27. Αυτές οι περιφέρειες είναι όλες στην Ευρώπη των 15. Καλύπτουν Βέλγιο, Ελλάδα, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε πολύ μεγάλο βαθμό και συγκεντρώνονται στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλέ από αυτές είναι περιφέρειες οι οποίες ποτέ δεν ήταν στη σύγκληση. Τέλος, οι υπόλοιπε περιφέρειες είναι στην ανταγωνιστικότητα και επασχόληση σε αυτήν την κατηγορία, στις πιο ανεπτυγμένες δηλαδή περιφερειές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτές που δεν θα στο μέλλον σε καμία περίπτωση ούτε στην σύγκληση ούτε στην μετάβαση. Ο πληθυσμός αυτός, αυτής της κατηγορίας, παραμένει λίγο πολύ ο ίδιος και βρίσκεται κατά κύριο λόγο, όπως θα περιμένει κανείς, στην Ευρώπη των 15. Δανία, Ιρλανδία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, οι κατοχώρες και η Σουηδία είναι 100% σε αυτήν την κατηγορία ανταγωνιστικότητα, δηλαδή οι πιο ανεπτυγμένε χώρες. Θα μπορούσα να σου πω και πολλά άλλα, υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία στη μελέτη, αλλά αυτά πολύ βασικά όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Τώρα, όσον αφορά την κατανομή της χρηματοδότησης, με ένα λόγια το ποιο παίρνει πόσα. Εδώ ε, έχουμε έναν πίνακα τον ο οποίος δεν φαίνεται δυστυχώς. Να σας πω όμως τα βασικά του χαρακτηριστικά. Οι προτάσεις της Κομισιόν προβλέπουν 336 δισεκατομμύρια στην συνοχή. Αυτό με μικρή μείωση, κατά λιγότερο από 5% των ποσών για τη συνοχή. Για δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, σύγκληση και συνοχή. Στην περίπτωση των ε, χωρών σύγκληση, έχουμε σημαντικέ μειώσεις κατά τον πέμπτο. Όμως σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε και αύξηση έως και 50%. Όπως και έχουμε αυξήσεις κατά ένα τρίτο για την εδαφική συνεργασία και για την ανταγωνιστικότητα σε συγκεκριμένες περιφέρειες, όπω και για την απασχόληση. Συν ένα πέμπτο. Αυτές οι μεγάλες αλλαγές στην κατανομή των πόρων αντικατοπτρίζουν και τις αλλαγές στην επιλεξιμότητα. Αν δείτε δηλαδή την ένταση των ενισχύσεων, δηλαδή την κατακεφαλήν καταβολή ενισχύσεων, αναπεριφέρεια, θα δείτε κάποιες επιμέρους διαφορές. Στις περιοχές που είναι ακόμα στη σύγκληση θα δείτε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι κατά κεφαλήν έχουμε αύξηση της χρηματοδότησης. Το ίδιο ισχύει σε κάποιο βαθμό για όσους είναι επιλέξιμοι για το Ταμείο Συνοχής. Όμως, στις μεταβατικές διατάξεις και πάντα για την κατακεφαλή χρηματοδότηση, εκεί τα κατακεφαλή ποσά θα πέσουν θεματικά. Από 100 ευρώ κατακεφαλή, που είναι αυτή τη στιγμή, σε περίπου 70 ευρώ. Κατακεφαλή και πάλι για τη νέα προγραμματική περίοδο η ένταση στις περιοχές ε, ανταγωνιστικότητας και είναι ενδιαφέρον αυτό, προτείνεται να αυξηθεί. Να αυξήσω την προσοχή σας επίσης ε, σε άλλες σημαντικές επιπτώσεις των προτάσεων της Κομισιόν. Όσον αφορά λέει το μηχανισμό της χρηματοδότησης. Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν τα ανώτατα όρια απορρόφησης, τα ανώτατα όρια συγχρηματοδότησης. Το μέγιστο της χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2,5% του ΑΕΠ. Πολύ διαφορετικό από το ανώτερο όριο για την παρούσα προγραμματική περίοδο. Αυτό το ανώτερο όριο, ως προς το ΑΕΠ δηλαδή, Μπορεί να ισχύσει. για το συγκεκριμένο έτος, χωρίς να την υπόψη δηλαδή η αύξηση του ΕΠ από χρόνο σε χρόνο. Αλλά αυτό είναι ακόμα συζήτηση. Όσον αφορά συνοχή και διαστατικά, είναι υποχρεωτική η κατανομή ενός τρίτου δύο τρίτων στην Ευρώπη των 12. Και επίσης δεν είναι σαφές ποια θα είναι η βάση για τον υπολογισμό των χρηματοδοτήσεων στις περιφέρειες σε μετάβαση. Υπάρχει, εκτιμάται τουλάχιστον ότι θα προκύψει ένα δίκτυο ασφαλείας για αυτούς που είναι τώρα στην σύγκληση και οι οποίοι θα χάσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας πάντως φαίνεται ότι τα δύο τρίτα του συνόλου των χρηματοδοτήσεων από την κατηγορία μετάβαση θα πάει στις παλιές ε, περιφέρειες και το 1 τρίτο σε περιοχές οι οποίες θα χρηματοδοτούνται όλο και λιγότερο. Τα είπα λίγο γρήγορα, αλλά ήθελα να σας πω ποια είναι τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τους υπολογισμού μας. Πιστεύω ότι θα άξει επίση εντάχει να σας πω ως προς τη μελέτη ότι περιγράφουμε τις παραμέτρους του διαλόγου που θα λάβει χώρα τους επόμενους μήνες ή και χρόνια. Οι θέσεις των χωρών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, πάντως από ό,τι βλέπουμε από τις δηλώσεις των χωρών μελών ως σήμερα, ο διάλογος θα αφορά καταρχήν το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για τη συνοχή, Ένα άλλο θέμα είναι το συνολικό ύψο του κοινοτικού προπολογισμού. Κάποιοι διαφωνούν επίση μετά για το πόσο το οποίο θα πάει στη συνοχή. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί. Άλλο δευτερεύον θέμα είναι η επιλεξιμότητα και η εσωτερική κατανομή πλέον των πόρων. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Κάποιοι λένε ότι όλοι πρέπει να είναι επιλέξιμοι, όλε οι χώρε πρέπει να είναι επιλέξιμε. Άλλε χώρες πιστεύουν ότι πρέπει τα πλουσιότερα κράτη-μέλη να μην χρηματοδοτούνται πλέον. Έχουμε επίσης και αυτήν τη νέα κατηγορία της μετάβασης, που είναι αρκετά αμφιλεγόμενη. Κάποια κράτη-μέλη την υποστηρίζουν, αλλά όμως ε, είναι ακριβώς κατά αυτής της δημιουργίας, της νέας κατηγορίας, γιατί θεωρούν ότι τα σχετικά όρια έχουν θεσπιστεί με τρόπο εντελώς αυθαίρετο και θα ήθελαν μια παραλλαγή μάλλον των phasing in και phasing out περιχών. Κάτι άλλο το οποίο δεν συζητήσαμε είναι το μερίδιο που θα πάει στο ΕΚΤΑ και στο ΕΤΠΑ και το κατά πόσον αυτό θα προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Παράλληλα όμως αυτό το έχουν απορρίψει πολλά κράτη-μέλη. Ύστερα υπάρχει ο χρηματοδοτικό μηχανισμός Connecting Europe, στο οποίο θα πάνε κάποια κονδύλια από τη συνοχή. Και αυτό προκάλεσε κάποιες αρνητικές απαντήσει από τις περιφέρειες, αλλά από και κράτη-μέλη, που φοβούν την τομεοποίηση της ε, πολιτικής αυτής, καθώς και την διαχείρισή της από το κέντρο. Αυτά όσον αφορά την γενικότερη πολιτική και τα χρηματοδοτικά. Όπως είπε ο συναδελφός μου, ο Δ. Μέντες θα σας πει λίγο περισσότερα για την έκθεση όσον αφορά το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό της μελλοντικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας δώσω επιγραμματικά μια εικόνα των βασικών στοιχείων για την πολιτική συνοχή. Βεβαίως ε, είναι πολυεπίπεδη, πολύ έχει διαστάσεις ε, και κοινωνικές και εδαφικές και περιφερειακές ε, που συνδέονται γενικότερα με στόχους ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και ως εργαλείο και μοχλός μπορούν να ειδωθούν σε τέτοιους καιρούς κρίσεις που βιώνουμε στη βιβλιογραφία βλέπουμε και επικρίσεις για τους στόχους ότι είναι συγκεχημένοι ή έχουν ε, κάπως οδηγηθεί σε κάποια συμφόρηση και περιπλοκή και χρειάζονται διευκρίνηση. Οι επικρίσεις αυτές δεν είναι τελείως ε, θεμητές, ούτε δικές. Είναι πολλές οι διαστάσεις και πολλές ε, πολιτικές και περιφερειακές και ε, εσωτερικές έχουν ε, και αυτές πολλές ε, πλευρές, πολλά επίπεδα και πολλές όψεις. Ε, βεβαίως Υπάρχει χώρος ε, για τη διευκρίνηση ε, των στόχων που επιδιώκουμε. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διαφόρων ε, επιπέδων, στρατηγικών, επιχειρησιακών και φιλοδοξιών. Να περιγράφονται καλύτερα οι στόχοι, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά και στο στάδιο του προγραμματισμού, να γίνεται διαφοροποίηση των στόχων από τους στόχους σηματοδότησης προς τακή ε, οδεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνηση ε, στο πώς ε, πληρούνται οι στόχοι ισότητας και αποτελεσματικότητας, όπως έλεγε και η ερεστική έκθεση, και τι γίνεται με τα ανταλλάγματα. Η εδαφική διάσταση, η περιφερειακή βεβαίως ενισχύεται, συστηματικοποιείται, στην πέμπτη έκθεση συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διάφορε ιδέες για την ενίσχυση της διάστασης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ε, μια πολύ ε, μεγάλη προσοχή στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, ε, φυσικές περιοχές, βιομηχανικές, ορεινές, αεροκατοικημένες κτλ. Αυτά γράφονται ρητά, αναφέρονται πλέον στη συνθήκη. Ε, γίνεται λόγος για ενίσχυση της αστικής διάστασης, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιμένει σε αυτό, αλλά και τη ε, λειτουργική διαχείριση και τελευταίο ενίσχυση της εδαφικής περιφερειακής συνεργασίας και οι λεγόμενες μακροπεριφέρειες. Τα κράτη-μέλη γενικά ήταν επιφυλακτικά απαντώντας την έκθεση συνοχής και τα περισσότερα στοιχεία για την ενίσχυση της αστικής διάστασης με ένα κατόφλι για προσημείωση ή ε, κάποιες ε, ειδικέ ρυθμίσεις για τις πόλεις και τα λοιπά. Ε, διαβάζοντας όμως τη βιβλιογραφία και μελετώντας το θέμα, ιδιαίτερα με αυτή τη λογική της εδαφικής συνοχής, Υπάρχει χώρος για περισσότερες εξειδικευμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει περισσότερη έμφαση στην ε, τοπική ανάπτυξη, στις τοπικές επενδύσεις ε, για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας ε, μεταξύ περιφερειών με πραγματικά διασυνοριακή σημασία και διεθνή άλλες στρατηγικές και επίσης θα πρέπει να είναι υποαίρεση η χρηματοδότηση σε σχέση ε, με την ε, γενικότερη ε, συνεργασία, με απλές διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία και στρατηγική καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με στρατηγικά έγγραφα, αλλά θα πρέπει και η ΕΣΠΟΝ που είναι το αντίστοιχο think tank να αξιοποιείται καλύτερα. Έρχομαι τώρα στη ε, στρατηγική συνοχή και τον προγραμματισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως πρότεινε ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για να ενσωματωθούν ε, τα διάφορα ταμεία διαχείρισης και με οριζόντιο συντονισμό, αλλά προτείνει και ε, καλύτερη και πιο στοχευμένη προσέγγιση μέσω συμβάσεων που είναι και δεσμευτικές ε, στα ε, διάφορα στρατηγικά προγράμματα ανάπτυξης ε, των κρατών, τα ΕΣΠΑ. Επίσης είναι και το θέμα που ενδιαφέρεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή για την κοινή στρατηγική μέσα σε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην εκπόνηση αυτών των θεμάτων. Υπάρχουν και διοικητικέ πτυχές για τις συμβάσεις εταιρικών ε, σχέσεων, βεβαίως τα κράτη-μέλη δεν θέλουν αυτό να είναι επιπλέον διαχειριστικό επίπεδο, έτσι, διοικητικό επίπεδο, που να μοιάζει κάπως με το προηγούμενο ε, πριν από δύο προγραμματικές περιόδους. Και η βασική ανησυχία επίσης και μέλημα είναι να μην υπάρχει υπερβαλλικός κατακαιρματισμός ε, ε, ε, των ενισχύσεων σε πάρα πολύ εξειδικευμένους κλάδους και τομείς. Επίσης τα νέα για τα διάφορα ταμεία και η διαφοροποίηση από κατόφλι σε κατόφλι για διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών και επενδυτικές προτεραιότητες. αποτελεσματικός έλεγχος και παρακολούθηση Συγγνώμη, πέρασα μια διαφάνεια. Ε, το πλαίσιο απόδοσης επιδόσεων είναι κάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εδώ είναι δύο τα βασικά στοιχεία, να υπάρχει μια σύνδεση, μια αιρεσιμότητα με κάποιους όρους ε, πριν και μετά την ενίσχυση ακούγονται διάφορες επικρίσεις και με δοθοδολογικού χαρακτήρα αλλά και ε, υπάρχει ένας κίνδυνος η πρόκληση ε, πώς να μην πολιτικοποιείται μια πολιτική να μην φορτίζεται πολιτικά δηλαδή μια ε, πολιτική ενισχύσεων να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και στην άμεση σύνδεση των μέσων με τη συνοχή. Ε, θα πρέπει εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις να ε, είναι περιορισμένοι σε αριθμό και να σέβονται την επικουρικότητα. Ποιε είναι οι προϋποθέσεις, αν θέλετε, τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση ε, της επιβολής αυτών των όρων υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και σημαντικές που φαίνονται και στη βιβλιογραφία. Χρειάζεται καλύτερη στόχευση στα προγράμματα, ε, ορισμός κοινών δικτών από την αρχή της προγραμματικής περίοδου. Επίσης, ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα σχέδια αξιολόγησης και να χρησιμοποιείται περισσότερη μελέτη αντικτύπου και πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μάλλον αποσιωπάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούσε να πει περισσότερα και να κάνει περισσότερα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρει πίν στη στρατηγική συζήτηση για το πώς μπορεί να τονωθεί αποτελεσματικότητα, δηλαδή να υπάρχει ένας πιο έντονος θεσμικός διάλογος και επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη πληροφορία για το Κοινοβούλιο και για άλλους ενεχομένους για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης. Προηγουμένως το ανέφερε ένας ε, Έλληνας Ευρωβουλευτής που είπε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ε, νωρίτερα διαθέσιμη, αλλά και Επίσης, οι εκθέσεις υλοποίησης και εφαρμογή θα πρέπει να δημοσιεύονται. Αυτό το καιρό πολλά κράτη-μέλη και πολλές περιφέρειες ε, δεν δημοσιεύουν καν αυτές τις εκθέσεις. Ε, ορισμένες ε, δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης. Αλλά είναι σημαντικό και για τη λογοδοσία, αλλά και για να βεβαιωνόμαστε ότι τα δεδομένα είναι ακριβώς υψηλής ποιότητος και τα στοιχεία. Και ένα τελευταίο, βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική μηχανή, όχι μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μπορεί να ανταποκρίνεται η διοίκηση. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας ε, απασχολήσει και στο μέλλον, αλλά αφορά τον εξυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών, τη μηχανογράφηση. Ε, σήμερα δίνεται μεγάλη ε, προσοχή στην κατάρτιση για καλύτερο σχεδιασμό, για καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων. βεβαίω και στην εφαρμογή και στην υλοποίηση τίθεται και ένα θέμα νομιμότητας όταν σύνονται αυτά τα συστήματα. η διαχείριση και το μοντέλο αυτό ε, γνώρισε πολλές επικρίσεις από τα κράτη-μέλη. Είναι πιεστικές οι προτεραιότητες, κυρίως να μην φορτώνονται τόσο πολύ ε, οι δικαιούχοι και ε, οι διαχειριστές με υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό είναι μεγάλη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζικές αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και αυτό προκύπτει από το δημοσιονομικό κανονισμό και από την ιδέα ας πούμε, που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο της γεωργίας για την πιστοποίηση, για την ετήσια καθάριση των λογαριασμών, για δηλώσεις ε, διαχειριστικές. Θα πρέπει να βρεθεί ε, η χρυσή τομή ε, για να συγκεραστούν οι προτάσεις με τις τρέχουσες πρακτικές το θέμα της αναλογικότητας. Ο έλεγχος και η διαχείριση θα πρέπει να είναι ε, αναλογικότερα του κινδύνου ή ε, του χρηματοδοτικού μεγέθους ενός έργου. Στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν διάφορες ε, ιδέες, αλλά Αυτό συζητείται, δηλαδή ε, όσο ε, χαμηλότερο είναι ο όγκος της χρηματοδότησης, τόσο χαλαρότερε θα πρέπει να είναι οι διαδικασίες. Αυτό ελέγχεται, γιατί μετά θα ακούσουμε επικρίσεις για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, η απλούστευση βεβαίως είναι μια προτεραιότητα πάγια για εναρμόνιση κανόνων επιλεξιμότητας, ε, για την ανάγκη να υπάρχει ένας συνολικότερος κανονισμός και να ε, απλουστεύονται και οι όροι και οι κανόνες για τις αποσμιώσεις με καταποκοπή ποσά. Αλλά δεν είμαστε βέβαια της άποψης ότι αυτό θα είναι πανάκια για να αντιμετωπιστεί η ε, πολυπλοκότητα και οι βαριές διοικητικές διαδικασίες. Προστιθέμενη αξία ολοκληρώνοντας. Βεβαίως και αυτό είναι περίπλοκο ζήτημα. Η έννοια και μόνο της προστιθέμενης αξίας καλύπτει ευρύ φάσμα ζητημάτων. Είναι και τα οικονομικά και η οικονομική προσθέμενη αξία της πολιτικής, αυτή η ε, ιδιότητα που να δρούν ως μοχλός, αλλά έχουν και άμεσες και έμεσες επιπτώσεις. Ε, για την οικονομική προσθετικότητα αυτό έχει και μεθολογικά προβλήματα. Πέρα από το γεγονός ότι κάθε δαπάνη είναι προσθετική. Πού θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Σε αυτή τη διάσταση της προστιθέμενης αξίας λόγω της πολιτικής. Σήμερα η προστιθέμενη αξία Ε, φαίνεται να συνδέεται με τις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 και ότι είναι ένας μηχανισμός για να φτάσουμε ε, σε αυτούς τους στόχους, στους ε, διάφορους τομείς, στα διάφορα κάθετα κανάλια διακυβέρνησης. αλλά πρέπει να οριστεί καλύτερα η προστιθέμενη αξία στην πολιτική. Βέβαια, ο κανονισμό λέγει ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι συμπληρωματική των εθνικών πολιτικών κτλ. Ωραία. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να το προωθεί. Από πλευρά ε, ε, των χρηματοοικονομικών μέσων, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι και στόχος της ε, ε, νομικής ασφάλειας και των διευκρινήσεων. Είναι δύσκολο αλλά αυτά να εφαρμοστούν στην πράξη. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πειραματίζεται περισσότερο με καινοτόμα προγράμματα και στο παρελθόν και πρωτοβουλίες επιτόπου στις περιφέρειες, αλλά σήμερα τίποτα δεν δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προχωρήσει με σένος και να πειραματιστεί. Βεβαίως θα πρέπει να θεωρηθεί και να προστευτεί ο κανόνας του νησιν 2 και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα. Και θα ήθελα να φέρω εδώ και μια βασική ε, επίκριση ότι αυτός ο κανόνας εμποδίζει ε, την ανάληψη κινδύνου και την καινοτομία. Αυτή η αρχή της εταιρικότητας έχει ατονίσει, έχει αυλυνθεί. Ίσως θα πρέπει να τονωθεί καλύτερα στον κανονισμό για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργεί στην πράξη, να υλοποιείται. Από την άλλη υπάρχουν και πιο ήπιες προτάσεις, ανταλλαγή εμπειριών, κάτι που ήδη συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα μπορούσε να έχει ε, μεγάλο αντίκτυπο και εδώ να δούμε πού εφαρμόζεται η αρχή της εταιρικής σχέσης ε, με σωστό τρόπο και στο πνεύμα που ε, διέπει τους κανονισμούς. Αυτά είναι μια επισκόπηση των βασικών στοιχείων της έκθεσης. Υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζω ότι έχουμε ζητήματα ε, πίεσης χρόνου. Με χαρά να ακούσω τα σχολεία σας και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Θα αρχίσει τώρα η συζήτηση. Ο Λάμπερτ Φαρνίστεροι έχει ήδη σηκώσει το χέρι του και θέλει το λόγο. Και ο Γιάννα Ορμπριχτ στη λίστα. Δεν ξέρω τώρα ποιο ζήτησε πρώτο το λόγο. Ο Λάμπερτ είναι πιο σημαντικό τέλεχο εδώ, έτσι δεν είναι. Όχι, απλώ θα μιλήσω πιο σύντομα. Στα αγγλικά ο κ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπειρογνώμονες ε, για τις επιδόσεις τους, γιατί την πρόλαβαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία μέρα νωρίτερα. Μπράβο, προλάβατε στο παραπέντε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ε, ενημερωτικά, εμπεριστατωμένα, μας δίνουν ε, πολλές ε, προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε την ίδια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με μελέτες και με σύγκριση των εμπειριών μας. Νομίζω βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά στις συζητήσεις μας και να οξύνουμε τις ιδέες μας. Έχω μία ερώτηση μόνο για το ε, Ευρώπη 2020. Μας ενδιαφέρει πολύ. Είπατε ότι θα είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ιδέα για το θέμα της Ευρώπης 2020. Μα αυτό είναι τρομακτικό. Είναι κρίσιμη στιγμή τώρα. Ε, ήδη δύο χρόνια ε, έχουμε αυτή την υπόθεση με ε, εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα λεγόμενα flagships. Τι είναι αυτά, μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε ή όχι. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την καινοτομία, σε όλες αυτές τις πολιτικές που έχουμε, τις πρωτοβουλίες αν δεν βλέπετε να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, μπορείτε να μας πείτε γιατί. Και φαντάζομαι ότι θα είναι ενδιαφέρουσε συζητήσει στο μέλλον. Ευχαριστώ, Γιάννη. Uh, Από όσο καταλαβαίνω, αυτή η συζήτηση αφορά την ε, συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει και λαμβάνει χώρα και όχι ε, δεν αφορά ακριβώς ε, την ε, συζήτηση για τον κανονισμό που θα κάνουμε αύριο. Στην ίδια την έκθεση που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κάνετε μια βαθιά ανάλυση και αναφέρεστε σε τέσσερα οράματα. Μόλις τώρα πήρα αυτό το υλικό και επομένως πραγματικά δεν μπορούσα να το μελετήσω εντελεχώς. Προσπαθώ να βρω μια, την απάντηση στο ερώτημα ποια από τα οράματα είναι το δικό σας όραμα, ποιο είναι αυτό που εσείς θεωρείτε καλύτερο και επίσης το άλλο ερώτημα, το, το όραμα που θεωρείτε καλύτερο ταυτίζεται με το όραμα της Επιτροπής. Εάν έχουμε τέσσερα οράματα, ποιο είναι το καλύτερο κατά την άποψή σας. Γιατί τα υπόλοιπα αφορούν τον αντίκτυπο. ή ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει, μπορεί να προκύψει ένα εξαιρετικό μείγμα διαφορετικών οραμάτων, ένα μείγμα διαφορετικής μεθοδολογίας, διαφορετικών τεχνικών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε την κρίση έτσι με έναν πιο οραματικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου την, το βέλτιστο όραμα. Και κάτι άλλο που ίσως αν διάβαζα προσεκτικά θα το έβρισκα στο κείμενο. Τι εννοείται ε, μακροπεριφέρειες, ε, τι, τι πιστεύετε για τις μακροπεριφέρειες ε, και την πολιτική που σχετίζεται με τις μακροπεριφέρειες. Πιστεύετε ότι είναι απόλυτα ξέχωρο από την διευθυντική πολιτική ή όχι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μονάχα για αποφάσεις ή για δηλώσεις. Στην ουσία μιλάμε για χρήματα. Επίσης, ε, διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων, ε, διακυβέρνηση έτσι όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, και ένα σχόλιο, εάν έχουμε αυτό το περιβόητο εργαλείο για την μεταφορά και εάν επιτευχθεί αυτή η μεταφορά χρημάτων από, την, από το Ταμείο Συνοχής, όχι απλώς να οριστούν τα χρήματα, αλλά να γίνει η μεταφορά των χρημάτων. Δεν θα έχουμε λοιπόν 2,5 αλλά σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικές χώρες θα έχουμε 2,5, σε άλλες χώρες 2,2, 2,1, 2,3. Αν ε, αυτή η κίνηση λοιπόν ε, του Επιτρόπου Μεταφορών ε, ευοδοθεί, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλες διαφορές γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να ε, ληφθούν ε, χρήματα και να μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ναι, η ερώτηση μου είναι εξή. Ε, καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για τη μελέτη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρόλαβα να τη δώσω τις λεπτομέρειές της, αλλά νομίζω θα μας βοηθήσει όλους. Η ερώτηση μου έχει ω εξή. Ασφαλώς ε, οι μελετητέ έχουν υπόψη τους τους στόχου της Ευρώπης 2020 και το γεγονό ότι εκεί υπάρχουν ε, πολιτικές και προτεραιότητες οι οποίες μπορούν να ελοπιθούν τόσο από τις περιοχές της σύγκληση, όσο και αυτές της ανταγωνιστικότητας όσο και της ενδιάμεσης. Ε, σε αυτή την αίθουσα και γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση η οποία λέει το εξής ότι για να επιτευχθεί ανάπτυξη, αν θέλετε για να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση, δεν είναι, και για να επιτευχθεί και μια σύγκληση βεβαίως, δεν είναι αρκετές οι πολιτικές της Ευρώπης 2020 και χρειάζονται και συμπληρωματικά μέτρα. Η ερώτησή μου στους μελετητές είναι η εξής. Από τη μελέτη τους βγαίνει το συμπέρασμα ότι εάν εφαρμοστούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020 πράγματι θα υπάρχει σύγκληση και σε τι βαθμό στο τέλος αυτής της πορείας. Μπορεί κανείς να το προσδιορίσει με έναν τρόπο σήμερα ή απλώς η όλη συζήτηση είναι στον αέρα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, μήπως μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα σχόλια και τις ερωτήσεις που έχουν ακουστεί. Ναι, είναι το πρώτο τμήμα των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω στην πρώτη και την τρίτη ερώτηση σχετικά με την Ευρώπη 2020. Ενδεχομένως υπερβάλαμε τις απόψεις των ε, κρατών μελών γιατί δεν προσπαθούμε να πούμε ότι η Ευρώπη 20, η 20 πολιτική συνοχής δηλαδή ε, δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την Ευρώπη 2020. Όντω πολλέ χώρε μέλη, κυρίως ε, ε, είναι πλουσιότερες θα καλωσορίσουν βεβαίως το πρόγραμμα την Ατζέντα 20, Ευρώπη 2020 γιατί ε, θα τους βοηθήσει να εστιάσουν καλύτερα στις ε, πολιτικές τους. Το ερώτημα είναι ο βαθμός στον οποίο ε, η Ευρώπη 2020 κατά πόσον θα χρησιμοποιήσει χρήματα από την ε, πολιτική συνοχή σε. κυρίως ε, ποια θα είναι η ανάλυση των διακυβευμάτων, των προκλήσεων ε, και σε επίπεδο κρατών μελών και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να οριστεί η βέλτιστη χρήση του Ταμείου Συνοχής, ε, η κατανομή των πόρων, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατανομή των πόρων. Ε, βεβαίως ε, κατανοούμε ότι ε, το earmarking κάποιων κονδυλίων βεβαίως είναι μια σαφής διαδικασία, κάνει ορατούς τους πόρους αυτούς. Αλλά πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε η Ευρώπη 2020 να μην μπει σε τρομερές λεπτομέρειες και ε, επίσης να μην υπάρξει υπερβολικός κατακαιρματισμός ή μάλλον υπερβολική θεωρητική αναφορά στους στόχους της ε, πολιτικής έτσι ώστε ανάμεσα στην εδαφική διάσταση και την, ε, και την υπερεθνική διάσταση να μην χάσουμε τους πραγματικούς στόχους. Um, Τώρα, το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει, να επιτευχθεί η σύγκληση. Ε, δίνεται μεγάλη έμφαση στην σύγκληση, στις προτάσεις, έτσι όπως τις αναγυγνώσκουμε εμείς. Επίσης, ε, ε, επικέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν. Ε, είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πολιτική συνοχής, η συνοχή και η σύγκληση, αυτά τα ζητήματα, να εξεκολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο του σκεπτικού οι ερωτήσεις που έθεσε ο Γιάνν Ορμπρεχτ. Δηλαδή ποιο είναι το όραμα το οποίο εμείς ε, στηρίζουμε. Στηρίζουμε πολύ την, ε, ε, το όραμα της Επιτροπής που βασίζεται στην εδαφική διάσταση. Εκεί που ενδεχομένως θα αποστασιοποιηθούμε λίγο είναι στο από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Ε, σχετικά με την ε, υλοποίηση προγραμμάτων ε, που θα πρέπει να γίνονται πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Ε, ίσως λοιπόν εμείς ε, να επιλέγαμε το bottom-up, τη διαδικασία από κάτω προς τα πάνω που λαμβάνει υπόψη ε, και τις υπάρχουσες δομές, τις περιφέρειες, Δεν φαντάζομαι, μάλλον νομίζω ότι ήδη και οι περιφέρειες τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα πρόσφατα. Επομένως, ε, καλό θα ήταν να δεσμευτεί η Κομισιόν ότι θα έχει μια ισχυρή διαδικασία διαδικασίας bottom-up. Ε, τέλος, είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά πιστεύω ότι ναι, υπάρχει δυναμικό ε, και αναφερόμενος στην κεντρική έκθεση ε, και λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της Επιτροπής, ε, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να δει, με, να αντιμετωπίσει με ευελιξία την εδαφική διάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές ε, γεωγραφίες ως βάση των νέων πολιτικών. και στην ουσία δηλαδή ας ξεκινήσει η διαδικασία να δούμε προς πώς θα πάει. Είναι ακόμα πάρα πολύ πρόημες αυτές οι εκτιμήσεις. Μπορούμε να μάθουμε από τις ε, εμπειρίες στην Βαλτική θάλασσα, στο Δούναβι. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε λίγο. Υπάρχουν όμως πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά αυτή την αντίληψη. Uh, Το μόνο που θα είχα να προσθέσω στην πρώτη ερώτηση για την Ευρώπη 2020 και πώς συνδέεται αυτό και την πληροφόρηση έχουμε. Οι ενσωματωμένες κατευθυντήριες γραμμές, οι ολοκληρωμένες μάλλον, εγκρίθηκαν πέρυσι και δόθηκε συνέχεια και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπουν ως υποσύνολο, ως θεματικές προτεραιότητες. Έχει γίνει και στο παρελθόν μια λίστα, ένας κατάλογος θεμάτων που είναι προτεραιότητες και βεβαίως είναι και ο προπολογισμό για το 2020 θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει με ειδικά κατόφια για την κλιματική αλλαγή, για την καινοτομία και για το ESF που είναι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει λοιπόν ε, πληροφόρηση και για την ανάπτυξη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν ε, διευκρινιστεί, μάλλον διευκρινίζει αυτό, ξεκαθαρίζει τι ακριβώς είναι το, η Ευρώπη 2020. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ γενικόλογο και καλύπτει τα πάντα. Υπάρχει όμως κάποια γενική καθοδήγηση, ένας προσανατολισμός και αύριο όταν εγκριθούν οι κανονισμοί θα έχουμε καλύτερη εικόνα αν θέλετε και μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Κύριε Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Εξαιρετικά επίκαιρη. Είναι καιρό να μιλήσουμε για τις κατευθυντήριε γραμμές, για την εφαρμογή τους. Φυσικά χρειάζονται σχετικοί πόροι. Το ερώτημά μου άφηνε ακριβώ αυτού. Γνωρίζουμε ότι η Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη. Πολλές φορές επερώμαστε γι' αυτό. Όμως, η αλληλεγγύη αυτή γίνεται και αντικείμενο αμφισβήτησης κυρίως εν ώψη του μέλλοντος, του μέλλοντος των χρηματοδοτήσεων. Υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχουν, υπάρχει εντύπωση ότι γίνονται διακρίσεις. Παράλληλα πρέπει να μειώσουμε τα χάσματα, τις διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Τώρα αν δούμε τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, τους μηχανισμούς στήριξης, όπως ας πούμε την συνοχή, και τα σχετικά κριτήρια, θα έλεγα ότι βλέπω, ας πούμε καταρχήν, ότι υπάρχει ένα τότε όριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως, όσο και αν φαίνεται αυτό λογικό και δίκαιο, αυτό θα θίξει τις λιγότερο ευνημένε περιοχές, τις φτωχότερες περιοχές. Ακριβώς επειδή εκεί το κρατικεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο. Ποιο είναι το σχολείο σα ω προ αυτό. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τελικά πώς, λειτουργεί, πώς λειτουργούν αυτοί οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Θα ήθελα να μου πείτε για την ελεγγύη και για την αρχή της μη, της, της μη μεταχείρισης. Λίσα Ρόλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πρόεδρος θέλει επίση το λόγο ε, για ερώτηση για σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει έχετε το λόγο. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον να ευχαριστήσω τον Τζον Μπάχλερ και την ομάδα του για την εξαιρετική αυτή μελέτη. Δεύτερον, να πω ότι πολλές από τις συστάσεις και τα συμπεράσματα συνάδουν και συμφωνούν με αυτά που έχουμε κάνει και εμείς. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά για τη μελέτη. Να διευκρινίσω ένα-δύο πράγματα που είπε ο Τζον στην αρχή όσον αφορά την αρχιτεκτονική της πολιτικής μας και τα στοιχεία σχετικά με την επιλεξιμότητα. Δεν θέλω να προδικάσω τους ε, υπολογισμούς που έχει κάνει ο καθένας, αλλά για τις διαφορετικές κατηγορίες και για το τι θα αλλάξει. Για την κατηγορία των, περι... των περιφερειών μετάβασης, εκεί θα έχουμε 51 περιφέρειες. Οι περισσότερες είναι εντός της Ευρώπης 15, Ας πούμε, στη Γαλλία έχουμε 10 περιφέρειες, στη Γερμανία 9, στο Βέλγιο 4, στη Φιλανδία 1, Ισπανία 4, Πορτογαλία 1, Πολωνία 1, Ηνωμένο Βασίλειο 9. Να, αυτή είναι, αυτή είναι κάποια νούμερα όσον αφορά την κατηγορία αυτή. Περιφερείς σε μετάβαση. Τώρα, όσον αφορά την κάλυψη αυτής της κατηγορίας, προφανώς αυτή είπαμε αντικαθιστά τις περιφερειές phase in και phase out. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκάλυψη 36,7 εκατομμύρια πληθυσμό, πάμε σε 72 εκατομμύρια για την περίοδο μετά το, 1900, το 2014. Και ανεβαίνουμε σε 51 από τις 27 σε 51 περιφέρειες με την καινούργια αυτή κατηγορία. Κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι η κάλυψη σε ή μάλλον η ένταση η κατακεφαλή ένταση της στήριξης. Στην Ευρώπη των 15 και στην Ευρώπη των 12 είχαμε τους σχετικούς υπολογισμού. Σήμερα για την Ευρώπη των 15 έχουμε 65 εκατομμύρια κατακεφαλήν το χρόνο. 65 ευρώ, να σχολείτε. Και αυτό αλλάζει σε 52 για την Ευρώπη των 15 και σε 264 για την Ευρώπη των 12. Βλέπουμε λοιπόν μια μικρή μείωση, αν θέλετε, για τα παλιά κρατημέλη και μια μικρή αύξηση για τα νέα. Και να διευκρινίσω αυτό που λέει η μελέτη για την αρχιτεκτονική και για την νέα κατηγορία. Όλα αυτά είναι απολύτως ακριβή. Τώρα κάποια νούμερα όμω μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις όσον αφορά την κάλυψη σε πληθυσμό και την κατακεφαλήν ε, ε, στήριξη καθώς και την κατανομή γενικότερα του προπολογισμού. Εκεί χρειάζεται λίγο να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Θα λέγαμε επίσης, ω προ όλα αυτά, ότι οι μελλοντικέ προτάσει θα συνοδευτούν και από μια μελέτη επιπτώσεων όπου θα αναλύνεται αναλυτικά και οι καλύψεις προς τον πληθυσμό και η κατακεφαλήν ένταση και η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού αλλά χώρα, περιφέρεια κλπ. Αυτά είναι προϊόν του σχετικού μοντέλου ανάλυσης. Οπότε δεν ήθελα να ρωτήσω κάτι, απλώς να διευκρίνησω αυτός προς τα νούμερα, ότι γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την μελέτη. Πρόκειται για εξαιρετικά επίκαιρη μελέτη ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συγγραφείς της. Κύριε Χομπλερ, χαιρόμαστε που χαίρεται η Κομισιόν. Δεν έγινε μόνο γι' αυτό η μελέτη <laughs> βεβαίω, αλλά ευχαριστούμε τη Μελισσά. Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι αν σε αυτό το πράγμα δεν είναι εξέλιξη ακόμη, ας ελπίσουμε ότι αυτά που θα δούμε αύριο δεν θα αλλάξουν πολύ, ειδικά για την νέα κατηγορία των, περιφερειών σε μετάβαση. Μια ερώτηση. Αναφέρατε όμω, και μάλλον δεν ξέρω ποιο το είπε, ίσω κάποιο από του δύο καθηγητέ, κάτι για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είπατε ενισχυμένο θεσμικό διάλογο, αν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμά, γιατί είμαστε ακριβώ στη φάση που συζητούμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνθήκης και στο πλαίσιο διαφορών πολιτικών. Είναι ένα από τα θέματα, ξέρετε, που προκύπτουν κάθε φορά που συζητούμε ε, το six το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της δημοσιονομικές προοπτικές και είναι κάτι που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όταν διαπραγματευόμαστε. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ε, πολιτική συνοχή, είναι ένα ερώτημα βάση, ε, στο πλαίσιο του νέου συστήματος. Εμείς έχουμε εξαιρετική συνεργασία εδώ και ένα μισό χρόνο με την Κομισιόν και πάμε πολύ καλύτερα για πρώτη φορά και με το Συμβούλιο. Οπότε ενισχύεται αυτός ο διάλογος. Εσείς όταν λέτε ο ρόλος μας στην πολιτική, τι έχετε στο μυαλό σας, αναζητούμε νέες ιδέες, αλλά αν έχετε κάποια ιδέα, πείτε μας. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το διάλογο αυτό που έχουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα. Από πολιτική απόψεω, κατά κύριο λόγο τουλάχιστον, το οποίο μου φέρνει στο μυαλό κάτι άλλο που συζητούσαμε πριν δύο μέρε, τότε δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο διάλογος για την πολιτική συνοχή και τα διευθυντικά ταμεία αποκτά μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν ασκείται το ελεγκτικό συνέδριο με την δήλωση εξυπηστία. Το λέω γιατί μας ενδιαφέρει και η αξιολόγηση αυτής της πολιτικής. Το πώς, αποτελεσματικά ξοδεύουμε τα κονδυλιά μας. Το ελληνικό συνέδριο φυσικά θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στο πώς η πολιτική αυτή προστατεύει τα συμφέροντα της Ένωσης και του προϋπολογισμού για να μην έχουμε απρόπτα, αλλά με την ευκαιρία της έκθεσης και του ελληνικού συνεδρίου θέλω να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση, ο διάλογος δεν έχει σχέση μόνο με αυτά. Καλό θέλει να συνδυάσουμε τον διάλογο αυτό με την αξιολόγηση που θα προτιμάσει η Κομισιόν. Ο διάλογος όμως θα έλεγα να είναι πιο εξορπημένος, να συγκεράζει όλες τις πτυχές αυτής της πολιτικής. Οπότε Καταθέτω αυτές τις ιδέες για συζήτηση. και για τους ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για γενικότερα δηλαδή προβληματισμό. Να δούμε. Αυτά είναι τα ερωτήματα, αυτά είναι τα ζητήματα αν θέλετε. Όχι για να μου απαντήσετε εδώ και τώρα, αλλά για περαιτέρω προβληματισμό, όπως είπα. Υπάρχει μια ερώτηση από εδώ. Παρακαλώ. Και αν θέλετε να πείτε κάτι και αυτό που λέει η Ελίζα. Okay, thank you. Um, ναι, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία θα ε θα έπρεπε να είχα επαναλάβει αυτό που λέει και η μελέτη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στα στοιχεία. Εμείς κάναμε την ανάλυση μας ε, λίγο μετά τη δημοσίευση της ατζέντα το 2020 και χρησιμοποίησαμε ε, τα στοιχεία του ΑΕΠ ε, κατά κεφαλή ε, του 2007-2008 τότε. Και για το 2009 δεν έχουμε στοιχεία, ακόμα για μερικούς μήνες δεν θα έχουμε. Και θεωρούμε ότι θα ήταν παραπλανητικό ή τουλάχιστον δεν θα έδινε την πλήρη εικόνα να δώσουμε τα στοιχεία μόνο από το 7 και το 8 διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον αντίκτυπο της κρίσης. Διάφορες χώρες επλήγησαν από την κρίση και σε κάποιο βαθμό έχουν εξέλθει ήδη με διαφορετικές ταχύτητες και αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε και νέα στοιχεία βάσει εκτιμήσεων και προβολών από εθνικές πηγές. Γι' αυτό έχουμε και κάποιες διαφορές με τα στοιχεία που ανέφερε προηγουμένως η Ελίζα Ρόλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα οριστικά στοιχεία που θα παραθέσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και ε, οπωσδήποτε θα ξανακοιτάξουμε και θα αναθεωρήσουμε τη δική μας ανάλυση και σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Μορκουνάιτε αναφερθήκαμε στο θέμα των οροφών είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπάρχουν διαφορές στο μηχανισμό Καταβολή των κονδυλίων, 2,5% του ΑΕΠ, έχει διαφορά από το 3,8% του ΑΕΠ, που είναι χώριο, άλλε φορέ είναι εθνικό το προϊόν ε, και δεν γίνονται υπολογισμοί με τον ίδιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία να επιστήσουμε την προσοχή ότι υπάρχουν διαφορές ενδεχομένως ανάλογα με τον τρόπο που υπολογίζονται όλα αυτά και οι χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί και όπως είπε και η Ελίζα Ρόλερ έχουμε και σύγκριση ε, της Ευρώπης των 15, των 12 αργότερα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων αυτών κρατών. Πάντως, ε, εμείς χτυπάμε καμπανάκια, προειδοποιούμε και την Επιτροπή σας για ζητήματα που πρέπει να μελετήσετε ή να προσέξετε. Βεβαίω θα σκεφτούμε τα όσα μας ε, προτείνει η καθηγήτρια κυρία Χιούμπνερ που θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ένα ρόλο στο διοργανικό διάλογο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προβολή των πολιτικών. Υπάρχει μια απογοήτευση κάθε χρόνο στη συζήτηση που γίνεται για τα σφάλματα, τους δείκτες σφαλμάτων. Θα ήταν πραγματικά ιδανικό ε, να συνοδεύεται και με μεγάλη προβολή της Επιτροπής σας όταν συζητάει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μόνο τα αρνητικά και τα σφάλματα. θα το ξανασκεφτούμε στο μέλλον λοιπόν ε, ε, πώς θα μπορεί να διατίθεται ε, αυτή η πληροφορία και τα στοιχεία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Μπάκλερ και τον κύριο Μέντες. Και ε, παρακαλώ να ε, ευχαριστήσετε και τη συνεργάτη σας και για την έγκαιρη κατάθεση της μελέτης και αν δεν διαφωνεί η Επιτροπή θα ζητήσω μια σύνοψη της μελέτης να δημοσιευθεί αύριο μαζί με το νομοθετικό πακέτο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελίσσα Ρόλερ για τα σχόλιά της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς να έχουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εκτιμούμε πάρα πολύ. και να ε, παίρνει και το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συνήθως ε, παρακολουθεί σιωπηρά ε, την παρουσίαση μελετών που αναθέτουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αποφάσεις από πλευράς Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μοιραστήκατε τις σκέψεις αυτές. Εδώ διακόπτεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο παρακαλώ οι συνάδελφοι όσοι φεύγετε τώρα φέρετε τις κάρτες σας. Μην ξεχάσετε γιατί έχουμε ψηφοφορίες.